Παρακαλώ πολύ, ας αρχίσουμε τις σημερινές μας εργασίες με τις ψηφοφορίες σε σχέση καταρχήν με την ε, μελλοντική προσχώρηση της Αλβανίας. Παρακαλώ καθίστε. Θα ήθελα να κάνουμε μία δοκιμή με τις κάρτες για να δούμε αν λειτουργούν και να δούμε βεβαίως και μήπως ε, ενδεχομένως κάποιος την ξέχασε. Λοιπόν, κάνουμε μία δοκιμή. Λοιπόν, χτυπήστε ένα κουμπί οποιοδήποτε, όποιο θέλετε. Αρχίζει η ψηφοφορία, η δοκιμαστική. Είμαστε 39, αλλά ψήφισαν 30. Ψήφισαν όμως μόνο 30 από τους 39 παρόντες. Έχετε πρόβλημα? Allora, l'onorevole Omaroiten ha l'apparecchiatura, possiamo mandare... Η κυρία Ομενρόιτεν έχει κάποιο πρόβλημα. Vabbè, manca ancora un sacco di gente. E a Brock? Buongiorno. Bene, allora... Υπάρχουν πολλοί που έβαλαν την κάρτα τους αλλά δεν ψήφισαν. Ah, Αρχίζουμε λοιπόν με το σχέδιο ψηφίσματος για την Αλβανία. Τροπολογία 8. Υπέρ παρακαλώ. Στην παράγραφο 1. Τροπολογία 8. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ. κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 20 λοιπόν, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 μέχρι τη λέξη δημοκρατικές εκλογές υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 σε δύο τμήματα υπέρ του πρώτου τμήματος υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίφθηκε δεύτερο τμήμα Θέλετε να ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε. Λοιπόν, αρχίζει η ψυχοφορία για το πρώτο τμήμα της 26. Ηλεκτρονική, η οποία και αρχίζει. 49... 50, 50 ψήφισαν. Κλείνουμε λοιπόν. 23 υπέρ 21 κατά. Δεύτερο, το δεύτερο ε, τμήμα καταπίπτει 27 υπέρ 27 κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1, η προφορική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 31 τώρα. Υπέρ. Ε, l'emendamento 29. Ε, Δεν ψηφίσαμε την 29. Ψηφίζουμε την 31. Υπέρ. Υπέρ Τη 31. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3. Συμβασμός 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 μόνο η λέξη πέτη 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά Ας κάνουμε έναν έλεγχο για την 52. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ονομαστική για την 51. Λοιπόν, κλείνουμε. 33-17 εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σωστά. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 55. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. 54 ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 54. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια να τα βλέπω γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει σωστή καταμέτρηση. Κλείνει η ψηφοφορία. 40 κατά 11. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59. Καταπίπτει 58, 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. 73 τώρα. 73 υπέρ παρακαλώ. Κατά Καλύτερα να ελέγξουμε. Την 73 αρχίζει η ονομαστική ψηφοφορία. 55 κάρτες ψήφισαν 52, 24 κατά 27 απορρίπτεται, 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται, 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά και πάλι πρέπει να ελέγξουμε 77 αρχίζει η ψηφοφορία 55 κάρτες έχουμε, ψήφισαν όμως 53. 31 υπέρ, 21 κατά. 22, 22 κατά. Εντάξει. Περνάει λοιπόν. 79, 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 92 προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93-94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 Ζητήθηκε έλεγχος για τις 93-94, αρχίζει η ονομαστική. Ψηφίζουμε επί των δύο 93 και 94. 53 ψήφισαν από τους 55, 28 κατά, 25 υπέρ, άρα απορρίπτεται. 95. Ναι, την ψηφίζουμε την 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε, αρχίζει η ονομαστική. Ψήφισαν 53-54 τώρα. 26 έναντι 25 εγκρίνεται για μία ψήφο. Για δύο, για δύο. Εν πάση περιπτώσει δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. 27-25. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 98 όχι, κατά πίπτη έχετε δίκιο. Συμβασμός 9 υπέρ. Κατά αποχές αεγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές εγώ θα έλεγα ότι απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 108. Α, όχι, καταπίπτει. 109. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω απορρίπτεται αλλά ας ελέγξουμε. 109 πρώτο τμήμα, αρχίζει η ψηφοφορία. «55 ψήφισαν από τους 57, κλείνει η ψηφοφορία, «33 υπέρ 22 κατά». Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 114 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τέσσερα. Τέσσερα Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. πέντε Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. έξι. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την ε, πρόταση ψηφίσματος αρχίζει η ψηφοφορία Αρχίζει η ψηφοφορία. Έχουμε 61, 61 ηλεκτρονικές κάρτες, αλλά ψήφισαν 60. 60 υπέρ, ένας κατά, καμία αποχή να συγχαρούμε τον εισηγητή. Ψηφίζουμε τώρα να συγχαρούμε, όπως είπα, τον εισηγητή και ψηφίζουμε τώρα την έκθεση για την διαδικασία προσχώρησης του Κωσυφοπεδίου. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σε δύο τμήματα η τροπολογία 31. Συγγνώμη, 3, 3 λέει ο πρόεδρος. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Είναι σαφές το αποτέλεσμα. 32-33 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 34 για τα διάφορα τμήματα. 34 ε, υπέρ. Κατά. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τη 34 που έχουν ενσωματωθεί όλες, όλα τα τμήματα. Ενιαία ψηφοφορία θα γίνει και για τα τρία τμήματα. Έχουμε 62 ψηφίσαντες, έκλεισε η ψηφοφορία, 26 υπέρ, 35 κατά. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγώ νομίζω ότι απορρίπτεται. Τι θέλετε να ελέγξουμε. 35. Αρχίζει η ψηφοφορία.

αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 δεν μπορώ να παρακολουθήσω διότι υπάρχει πρόβλημα με, την, με τον κατάλογο του ΕΛΚ. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ψηφοφορία γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με τον κατάλογό μας. Ε, <laughs> ε, Η δική μας λίστα έχει ένα πρόβλημα. Να συγκεντρωθείτε και να ησυχάσετε. Εν πάση περιπτώσει, αντίχειρας πάνω, αντίχειρα κάτω, όπως θέλετε. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42. Ψηφίζουμε μαζί όλα τα τμήματα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43. Και εδώ έχουν ενσωματωθεί τα διάφορα τμήματα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είμαι σίγουρος ότι έχει απορριφθεί, άρα ας αρχίσουμε την ονομαστική για την 45. Εδώ βλέπω δύο τμήματα, λέει ο πρόεδρος. Όχι, όχι, είναι ενιαία. 62 ψήφισαν, Κλείνει η ψηφοφορία. 33 κατά 29. Περνάει. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 49 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά νομίζω πρέπει να ελέγξουμε 49 πρώτο τμήμα αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ε? για το πρώτο τμήμα του 49 ψήφισαν 63 34 κατά 28 υπέρ. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51. Και εδώ είναι ενιαία η ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 52-53 υπέρ κατά δεν είναι σαφές ελέγχουμε ηλεκτρονικά τις 52-53 παρακαλώ ψηφίστε τώρα Έχουμε 64 κάρτες, καρτέλες αλλά 62 ψήφισαν. Οι 22 κατά 31 υπέρ. Περνάει. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56. 56. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 Ενιά ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 61 ενιαία ψηφοφορία όλων των τμήματων υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε? Ας ελέγξουμε.

κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίφθηκε συγγνώμη συγγνώμη με συγχωρείτε εκφράστηκα λάθος απορρίφθηκε 67. Για την 66 ζητήθηκε έλεγχος. Ελέγχουμε. Για την 66. 66. 66. Ελέγχουμε. 63 ε, ψήφισαν, 44 κατά, 19 υπέρ απορρίφθηκε. 67 υπέρ, κατά, απόχες εγκρίθηκε. 68 υπέρ, κατά, απόχες εγκρίθηκε. 69 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίφθηκε. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 73 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 74 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 75 και 106 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα δεύτερο τμήμα ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις 75-106 από κοινού. 64 ε, κάρτες, αλλά ψήφισαν 61, 62. Κλείνει η ψηφοφορία. 20, 28 ε, υπέρ, 34 κατά. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 80 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Την 86 αρχίζει η ψηφοφορία. Έχουμε 63 ψηφίσαντες. Κλείνει η ψηφοφορία 33 υπέρ 30 κατά. Εγκρίνεται. 87 υπέρ Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Καταπίπτουν αυτές οι τρεις. Άρα πάμε στην 89. 89. Ενία ψηφοφορία των διαφόρων τμήματων υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ, όχι έκανα λάθος λέει ο πρόεδρος, εγκρίναμε την 113, άρα καταπίπτει 115-116 υπέρ, υπέρ της 116 κατά, αποχές απορρίπτεται 117, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ της 117 πάντα. Κατά αποχές νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Θέλετε να ελέγξουμε όμως. Λοιπόν, δεύτερο τμήμα της 117. Αρχίζει η ψηφοφορία. 64 καρτέλες, 62 ψήφισαν, κλείνει η ψηφοφορία, 40 υπέρ, 20 κατά. Δεν είχατε σηκώσει σωστά τα χέρια. Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται καταπίπτει, αποσύρθηκε μάλλον 120, 121 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται η προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 100, ε, επί της 123. Αρχίζει η ψηφοφορία. ...62 ψήφισαν, οι 28 κατά 34 υπέρ εγκρίνεται, 124 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 125 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 128 δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, Απορρίπτεται, με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρος. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε δεύτερο τμήμα της 128. Ονομαστική. ...63 ψήφισαν, από τους 64, 22 κατά 41 υπέρ, εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 μαζί με 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αποσύρεται 139-140, πάμε στην 141 υπέρ κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να ελέγξουμε. 141 ελέγχουμε. 63 ψήφισαν, πέρας 17 κατά 45 υπέρ. Μεγάλη πλειοψηφία, αλλά δεν την έβλεπα με τα χέρια. Περνάει. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ. Ηλεκτρονική επί της 142 ζητήθηκε. 142 ψηφίζουμε. 63 ψήφισαν, πέρας, 40 κατά, 23 υπέρ. Απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ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 αν θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε την 149. ...62 ψήφισαν από τους 64, 33 κατά, 28 υπέρ, 34 κατά, άρα απορρίπτεται 150 υπέρ. Κατά, Αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 153, 54 και 55. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 156 Μα ήταν σαφές. 153, 54, 55 θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε για τις τρεις. 64 καρτέλες έχουμε, αλλά 61 ε, ψήφισαν, 42 κατά, 18 υπέρ, όπως βλέπετε απορρίφθηκαν. 156. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ κατά Όχι, καταπίπτει. Εγκρίναμε την 136. Άρα καταπίπτει 161, με συγχωρείτε. Άρα έχουμε 162, 163, 164 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 165. Ξεχωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα στο προήμιο α17 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 20. Εγκρίναμε την 19, όχι, απορρίφθηκε, άρα ψηφίζουμε την 20, 20 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 22. Μάλλον για την 21 ζητήθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία και αρχίζει. Ήταν σαφές αλλά για μερικούς δεν ήταν. Λοιπόν, 21. Χρειάζεται και ο έλεγχος καμιά φορά πέρας 46 κατά 12 υπέρ απορρίφθηκε 22 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. «26. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά γιατί μάλλον εγκρίνεται». «63 σεσάντα 62...» ψήφισαν 62 πέρας, 16 κατά 42 υπέρ. Εγκρίνεται λοιπόν. 26 υπέρ. Α, όχι, αυτή ψηφίσαμε. Συγγνώμη, 27, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά απορρίπτεται 28 υπέρ κατά μάλλον να ελέγξουμε 28 αρχίζει η ονομαστική ψηφοφορία ελέγχουμε 63 καρτέλες αλλά ψήφισαν 61 πέρας 34-27 εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε καλύτερα. Ελέγχουμε για την 2. ...62 ψηφίσαντες, 27 κατά 33 υπέρ εγκρίθηκε. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5, 6 αποσύρονται, 7, 8 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται, ξεχωριστά τμήματα για την 9, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε καλύτερα, πρώτο τμήμα της 9, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 61 ε, ψήφισαν. 28-28 ισοψηφία. 29 ε, είναι υπέρ. Δεύτερο τμήμα της 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγώ νομίζω ότι έχει εγκριθεί 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15-16 Με συγχωρείτε, έκανα εγώ λάθος. Εγκρίθηκε. Εγώ έκανα λάθος, λέει ο πρόεδρος. 15-16 από κοινού υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την πρόταση στην τελική της μορφή. Αρχίζει η ψηφοφορία. 61 ψήφισαν, 63 καρτέλες έχουμε όμως, κλείνει η ψηφοφορία. 46 υπέρ, 14 κατά. Να συγχαρούμε τον εισηγητή, εγκρίθηκε. Passiamo alla votazione. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για την Ισλανδία. Προφορική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Καταπίπτει 16-17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ Κατά. Καλύτερα να ελέγξουμε, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. 21 αρχίζει η ψυχοφορία Ε, 57 ψήφισαν ηλεκτρονικά. 34 κατά, 22 υπέρ, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεν συμφωνείτε? Ωραία, ας ελέγξουμε. Αρχίζουμε τον έλεγχο για το συμβασμό 3 δεύτερο τμήμα. Έχουμε 59 καρτέλες, 56 ψήφισαν, κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 30 κατά, 26 υπέρ. 31. γιατί το δεύτερο τμήμα της 3 απορρίφθηκε. Ωραία, ψηφίζουμε την 31. Όχι, όχι, έκανα λάθος. Ψηφίζουμε... 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμό 4 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίθηκε. Συμβασμός 5 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίθηκε. Συμβασμός 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 45 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίφθηκε. Ε, 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμός 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο 2, μπροκ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά,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 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική, μάλλον ένα, ένα υπέρ. Όχι, καταπίπτει. Έχει εγκριθεί η προφορική. Άρα περνάμε στην προφορική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά για την πρόταση στο σύνολό της. Αρχίζει η ψηφοφορία. Έχουμε 56 καρτέλες. 54 ψήφισαν. Πέρας. 53 υπέρ, 1 κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Εγκρίνεται η πρόταση ψηφίσματος. Τελευταία ψηφοφορία Προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης. Αποσύρεται η 1 και 3, άρα προφορική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2. Προφορική. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 7. Προπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά Α, με συγχωρείτε, ε, ναι. Ε, έκανα λάθος, λέει ο πρόεδρος. 9. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την πρόταση στο σύνολό της. «56 καρτέλες έχουμε, 53 ψήφισαν και η κυρία Μενρόιτεν Απλώς να σας πω ότι αρχίσαμε εγκαίρος και τα καταφέρατε πολύ καλά. Να σας συγχαρώ λοιπόν. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίο αυτό το χάιδεμα από μια τέτοια κυρία. Λοιπόν, 41 3 κατά 4 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Να διακόψουμε για λίγα λεπτά. Σε τρία λεπτά ξαναρχίζουμε.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 possiamo. sta ancora telefonando. C'è un po' di confusione. And not the Madrid version. I mean the council version. The council version of the. yeah, so I can propose the 3rd of May version. As, I, I like the, the, the first. Uh,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 Ehm, Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε τώρα για να αρχίσουμε την ακρόαση του δόκτωρος Μιγκαρέλη αναπληρωματικού διευθυντού για τις σχέσεις με το Μαγρέμπ και γενικότερα της Μεσογειακής Λεκάνης που θα μας μιλήσει σήμερα για την εξέλιξη των σχέσεων αυτών, των ιδιότυπων σχέσεών μας με τη Λιβύη. Γιατί όπως γνωρίζετε δεν συμμετέχει στους μηχανισμούς της πολιτικής καλής γειτονίας και θα συνεχίσουμε σήμερα αυτά που είχαμε συζητήσει από το 8 ήδη. Περιοδικά μας πληροφορούν και πρέπει να είμαστε πληροφορημένοι και ενημερωμένοι για την εξέλιξη των σχέσεων. Γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε από κοινού την ευθύνη του θέματος αυτού. Παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και θα θέλαμε, θα θέλαμε λέγω, να υπάρξει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη Λιβύη. Ευχαριστώ τον συνάδελφο παντέρη που οργάνωσε τη συνάντηση αυτή. Είναι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγρέμπ. Ehm, e ε. Ας μην χάσουμε άλλο χρόνο. Αρχίζουμε τη συζήτηση και την ακρόαση και δίνουμε αμέσως το λόγο στον κύριο και δόκτορα Μιγκαρέλη. Κύριε Πρόεδρε, για τέταρτη φορά μου δίνετε τη δυνατότητα να σας αναφέρω την εξέλιξη των σχέσεων Ένωσης και Λιβύης και σας ευχαριστώ γι' αυτό καθώς και για την πρόσκληση των συναδέλφων μου για να δούμε από κοινού ποιες είναι οι πρόοδοι αλλά και οι δυσκολίες. Βεβαίως καθ' όλες τις διαπραγματεύσεις είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώνουμε και να σας γνωστοποιούμε τις δυσκολίες που τυχόν υπάρξουν ώστε να δούμε από κοινού ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων και όλα αυτά βέβαια σύμφωνα με το άρθρο 218 της συνθήκης που απαιτεί από την Κομισιόν να εφαρμόζει ως το δυνατόν να συνδυάζει και το Κοινοβούλιο τις διαπραγματεύσεις αυτές. Υπάρχει η Συμφωνία Πλαίσιο του Συμβουλίου του Ιουλίου 2008 και βάσει αυτής αρχίσαμε τον Νοέμβριο του 2008 τις διαπραγματεύσεις. Από τότε μέχρι τον Ιούνιο σήμερα, φέτος, 7 συναντήσεις οργανώθηκαν, πότε στη Λιβύη, πότε στις Βρυξέλλες. Πότε στην Τρίπολη, πότε στις Βρυξέλλες και η τελευταία έγινε πρόσφατα στην Τρίπολη. Πού βρίσκονται λοιπόν τα πράγματα. Μέχρι τώρα μπορέσαμε να κλείσουμε προσωρινά τρεις τίτλους της μελλοντική συμφωνίας. Οι τρεις αυτοί τίτλοι επί τους οποίους υπάρχει προσωρινή συμφωνία είναι οι γενικές αρχές των σχέσεων, η χρηματική συνεργασία, δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους, με τι εργαλεία μάλλον θα μπορέσουμε να κατορθώσουμε να εφαρμόσουμε την συνεργασία αυτή τεχνικά και τέλος τα γενικά θεσμικά θέματα. Συμφωνήσαμε επί της γενικής θεσμικής αρχιτεκτονικής της μελλοντικής συμφωνίας με λίγα λόγια και γι' αυτό προσωρινά κλείσαμε αυτά, αυτούς τους τίτλους. Κατά τη διάρκεια της 7ης συνάντησης διαπραγματευθήκαμε όλα αυτά τα θέματα εκτός από τα τρία που ανέφερα καθώς και το θέμα του εμπορίου και των συναλλαγών γενικότερα που δεν μπορέσαμε ακόμη να εγκρίνουμε κείμενο να υποβάλουμε κείμενο στους συναδέλφους μας από την Λιβύη. Για όλα τα θέματα λοιπόν που πραγματευτήκαμε στη Λιβύη έγιναν σημαντικές πρόοδοι ιδιαίτερα στα θέματα του πολιτικού διαλόγου της οικονομικής συνεργασίας και της τομεακής συνεργασίας. Το θέμα που υπήρξε το πιο αμφιλεγόμενο και το πιο δύσκολο ήταν το εμπόριο προφανώς και λέω προφανώς καταρχήν γιατί αυτό είναι γνωστό πρόβλημα. Ξέρετε ότι τα εμπορικά τμήματα της συμφωνίας ε, υπήρξαν ιδιαίτερα δύσκολα στη συζήτηση και επίσης προσθέτω προφανώς διότι σχεδόν όλες οι συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε με τρίτες χώρες όπως τη Ρωσία, την Ουκρανία, τις χώρες του Καυκάσου στο μέλλον, τη Συρία, με την οποία υπογρά... καταλήξαμε τις διαπραγματεύσεις αλλά δεν υπογράψαμε ακόμη τη συνθήκη, το Ιράκ, όπου επίσης δεν έχει υπογραφεί ακόμη η συμφωνία. Σε όλες αυτές τις συμφωνίες το πιο δύσκολο θέμα ήταν πάντοτε το εμπορικό. Για τον πολιτικό διάλογο οι Λίβοι εταίροι μας υπήρξαν πολύ ανοιχτοί, εισήκουσαν τα αιτήματά μας και τις συστάσεις μας. Πράγμα που μας επιτρέπει να είμαστε σχεδόν σε τελική φάση των διαπραγματεύσεων και για αυτό το θέμα. Η Λιβύη δέχτηκε να υπάρξει διάλογος και για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θέμα που επί χρόνια προσπαθούμε να το θέσουμε με όλους μας τους εταίρους. Στις αρχές των διαπραγματεύσεων δεν ήταν προφανές ότι θα έχονταν οι Λίβοι, αλλά το δέχτηκαν. Δέχτηκαν δηλαδή να υπάρξει διάλογος και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ή τον εκδημοκρατισμό. Επίσης δέχτηκαν τις προτάσεις μας για την καταπολέμηση, για την καταστροφή των όπλων μαζικής καταστροφής ακριβώς και την ε, ρήτρα που βάζουμε πάντοτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και που γενικά λέει ότι τα συμβαλώμενα μέρη μπορούν να αναστείλουν τη συμφωνία αν διαπιστώσουν ότι η άλλη πλευρά δεν σέβεται τα δικαιώματα και τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Εύκολο είναι να γίνει δεκτή αυτή η ρήτρα, πολύ πιο δύσκολο να εφαρμοστεί. Έχουμε πρόσφατα, πρόσφατα ενθυμήματα για τέτοια προβλήματα, όχι με τη Λιβύη. Σοβαρό πρόβλημα αποτέλεσε το αίτημά μας να μπει στη συμφωνία και μία παραπομπή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο γιατί μας είπαν πολλές φορές ότι δεν έχουν δεχτεί, δεν έχουν συνυπογράψει το καθεστώς της Ρώμης και ούτε έχουν την πρόθεση να το πράξουν. Γι' αυτό θελήσαμε να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός σύμφωνα με τον οποίο να δεχτούν να γίνει παραπομπή στο ότι είναι απαράδεκτη η ατιμορρησία που παρατηρείται για εγκλήματα που θεωρούνται ιδιαίτερως ιδεχθεί από τη διεθνή κοινότητα, δηλαδή γενοκτονίες, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος. Επαναλαμβάνω, ζητήσαμε να μπει στο κείμενο της συμφωνίας κάποια παραπομπή στην κοινή μας δέσμευση, Ένωση και Λιβύη, ώστε τα σοβαρότερα εγκλήματα που δέχεται ως τέτοια η διεθνής κοινότητα να μην παραμένουν ατιμόρυτα. προς στιγμή είναι ο μόνος συμβιβασμός επί του οποίου ίσως μπορέσουμε να καταλήξουμε. Μας δήλωσαν όμως αρχιτά ότι η αναφορά η παραπομπή στο διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο και στο καθεστώς της Ρώμης για αυτούς είναι απαράδεκτη και αδιαπραγμάτευτη. Και δεν είναι οι μόνοι που μας λένε κάτι τέτοιο. στι συμφωνίε που διαμορφωνόμαστε με τρίτες χώρες, πολλές από αυτές, μερικές από τις οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντική οι εμπορικοί εταίροι μα, αρνούνται να γίνει ακόμη και μια απλή παραπομπή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κατά τα άλλα για τον πολιτικό διάλογο υπάρχει συμφωνία εφόλων των θεμάτων. Και αυτό δεν είναι και μικρή επιτυχία. Για την μετανάστευση παραμένουν ακόμη πολλά εκρεμή σημεία. Το πρώτο είναι βέβαια η επανεισδοχή των παρανόμων μεταναστών που δεν είναι μεν πολίτες της Λιβύης αλλά έχουν περάσει από τη Λιβύη. Δηλαδή προσπαθούμε πάντοτε με τρίτες χώρες ιδίω γειτονικέ να έχουμε τέτοιες συμφωνίες επανεισδοχής κατά τις οποίες οι τρίτες αυτές χώρες δέχονται γενικά σχετικά εύκολα να πάρουν πίσω στις, τους παράνομους μετανάστες που έχουν συλληφθεί στην Ένωση αλλά που έχουν περάσει από τη χώρα αυτή. Οι Λίβοι δεν δέχονται πολύ εύκολα να δεχτούν να επιστραφούν οι παράνομοι μετανάστες που έχουν συλληφθεί στην Ένωση. Αλλά θα ήταν πράγματι δύσκολο να δεχτούν να πάρουν στη Λιβύη όλους τους δυστυχείς παράνομους μετανάστες από την Αφρική που περνώντας από τη Λιβύη έχουν φτάσει μέχρι την επικράτεια της Ένωσης. Μας είπαν ότι και για αυτούς είναι αδιαπραγμάτευτο το, και, για, και αυτό το θέμα είναι αδιαπραγμάτευτο για αυτούς. Εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια έχουμε όμως τέτοια συμφωνία με το Μαρόκο αλλά δύσκολη και αυτή. Και σας επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Λιβύης ότι δεν δέχεται εύκολα αυτή τη ρήτρα. Οι περισσότεροι εταίροι μας δεν τη δέχονται. Άλλο δύσκολο θέμα και κρεμές για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι το θέμα της μεταχείρισης των αιτητών ασύλου. Εμείς επιμένουμε η Λιβύη να διασφαλίζει την προστασία όσων ζητούν πολιτικό άσυλο και να εφαρμόζουν την αρχή της μη έκδοσης. Αλλά η δυσκολία είναι ότι η Λιβύη δεν έχει συνυπογράψει τη συνθήκη της Γενέβης του 51 και μας είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να το πράξει σύντομα. Και άρα δεν θέλει να γίνεται παραπομπή ούτε σε αυτή τη συμφωνία, Επίσης, είναι και αυτό μια πραγματική δυσκολία γιατί για μας εμείς θα θέλαμε μέσω της υπογραφής αυτής της συμφωνίας πλαισίου να υπάρξει κάποια πρόοδος και για την προστασία των αιτητών εσύλου και των προσφύγων από τη Λιβύη γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί και εδώ έχει παγώσει το θέμα και προσπαθούμε να βρούμε κάποιον συμβιβασμό. Πρέπει επίσης να σας πω ότι η Λιβύη δέχτηκε παρόλα αυτά να γίνει παραπομπή στην αρχή της μη έκδοσης μεταναστών που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Δηλαδή δεν αναγνωρίζουν μεν την έννοια του πρόσφυγα, αλλά δέχονται να γίνει παραπομπή στην αναγκαιότητα να μην εκδίδονται οι μετανάστες που χρειάζονται διεθνή προστασία. Έγινε ένα βήμα λοιπόν δεν ε, έγινε ακόμη δεκτό αυτό που θέλαμε, αυτό που προβλέπει η εντολή μας, αλλά παρόλα αυτά έγινε ένα βήμα. Βεβαίως στα πλαίσια της πολιτικής θεωρήσεων και μετανάστευσης η Λίβοι όπως και οι άλλοι εταίροι μας ζητούν συμφωνία για να διευκολυνθεί η χορήγηση θεωρήσεων για τη διαμονή ορισμένων κατηγοριών Λιβύων πολιτών βραχυπρόθεσμη στην Ένωση αλλά εδώ δεν έχουμε την εντολή των κρατών μελών να συμπεριληφθεί μια τέτοια ρήτρα στη συμφωνία. Τέλος υπάρχει το εμπορικό όπου καθώς σας είπα πολύ μακράν από συμφωνία είμαστε. Οι συνάδελφοί μας που διαπραγματεύονται το θέμα αυτό μας λένε ότι πρώτον η Λιβύη δεν έχει πολλές διεθνείς εμπορικές συναλλαγές λόγω της κλειστής της οικονομίας και γι' αυτό έχει δυσκολία να μιλήσει τη συνήθη εμπορική διεθνή γλώσσα. Δηλαδή με βάση τις εμπορικές συμφωνίες πρέπει να τους τα εξηγήσουμε όλα για να τα καταλάβουν. Αρχίζουμε από το μηδέν. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος λοιπόν από ότι με τους εταίρους μας που ήδη γνωρίζουν τα ιωθώτα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Και είναι και αυτό αρκετά τεχνικό θέμα και πρόβλημα. Δεύτερον, θα θέλαμε να υπάρξει σαφής δέσμευση της Λισβής να δεχτεί τις αρχές του ΠΟΕ. Και εδώ υπάρχει δισταγμός εκ μέρους της Λιβύης. Επίσης δυσκολία, δυσκολευόμαστε να τους κάνουμε να δεχτούν τη ρήτρα του παγώματος standstill κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, να μην αυξήσουν δηλαδή τους δασμούς τους όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Και αυτό είναι βασική αρχή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, αλλά για τους Λίβιους είναι κάτι καινούργιο και όχι προφανές. Τέλος, εξετάζουν αυτή τη στιγμή, επανεξετάζουν την οικονομική τους νομοθεσία, κυρίως τους δασμούς, και διστάζουν και επ' αυτού να την αλλάξουν. Εδώ είναι μια πραγματική δυσκολία λοιπόν στα εμπορικά θέματα και οι συνάδελφοί μας που τα διαπραγματεύονται σκέφτονται αυτή τη στιγμή ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να τα παρουσιάσουν όλα αυτά στους Λίβιους. Θα οργανώσουμε σεμινάρια στις Βρυξέλλες μέσω του ΤΑΓΕΞ για να εξοικειωθούν οι Λίβοι συνάδελφοί μας με το κοινοτικό εκτιμένο σε ορισμένους τομείς και επίσης οργανώνουμε πολλές τεχνικές συναντήσεις μεταξύ των δύο, μεταξύ δύο επισήμων συναντήσεων για τις διαπραγματεύσεις γιατί το ζήτησαν επανειλημμένως οι εταίροι μας ότι θέλουν οι διαπραγματεύσεις να λήξουν, να καταλήξουν ή δυνατόν μέχρι το τέλος του χρόνου, αύριο δηλαδή. Αν μπορέσουμε να οργανώσουμε τρεις ακόμη διαπραγματευτικές συναντήσεις το Σεπτέμβριο, μέσα Νοεμβρίου και το Δεκέμβριο, ίσως τότε να μπορέσουμε να καταλήξουμε, να λήξουμε τις διαπραγματεύσεις για τα κυριότερα θέματα που παραμένουν ακόμη εκκρεμοί. Αλλά θα ήθελα να επιμείνω ότι υπάρχουν ακόμη μερικά πολιτικά προβλήματα που τα θεωρούν αδιαπραγμάτευτα και ασάφεια μεγάλη ως προς το τι θα γίνει στα εμπορικά. Ιδού η σύνοψη που θα μπορούσα να σας κάνω για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Καταλήγω λέγοντας ότι θεωρούμε σημαντικό να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις ακόμη και αν δεν πετύχουμε όλα μας τα θέματα, διότι μέσω μιας τέτοιας συμφωνίας θα είχαμε μια θεσμική βάση για να υπάρξει τακτικός διάλογο σε όλα τα επίπεδα με εταίρους με τους οποίους έχουμε ορισμένα κοινά συμφέροντα, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ας πούμε, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τα ενεργειακά και άλλα, και με τους οποίους από την άλλη έχουμε και διαφορές. Αν καθοριστούν οι γενικότερες θεσμικές τα γενικότερα θεσμικά πλαίσια ενός τέτοιου διαλόγου θα μπορούσαμε τότε τακτικότερα και εφόλων των επιπέδων και θεμάτων να τα ξανασυζητούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Δόκτωρα Μιγκαρέλη, δίνουμε το λόγο στην κυρία ε, Γκόμες, η οποία είναι η συγγήτρια της ΑΦΕΤ ως προς τη συμφωνία με τη Λιβύη. Σας ευχαριστώ κύριε Μιγκαρέλη για την εισήγησή σας. Euh, Θα ήθελα να σας ρωτήσω, να σας υποβάλω μάλλον μία ερώτηση. Ποια είναι η νομική βάση αυτής της διαπραγμάτευσης. Ξέρουμε για την εντολή, αλλά αναμένουμε τη νομική βάση. Και Χαίρομαι για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί, όμως καταγράφω αυτά που μας είπατε, ότι δηλαδή ότι δεν έχει επιληθεί το ζήτημα της ε, μνήας ή της ε, παραπομπής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ίσως ε, γίνει ειδική μνήα στην αποδοχή της, στη μία αποδοχή της ατιμορρησίας για τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει ως προς τη μετανάστευση και τη χορήγηση πολιτικού ασύλου. Γνωρίζουμε ότι η Λιβύη ποτέ δεν κύρωσε την ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες του 1951 και ίσως επέλθει συμβιβασμός σε σχέση με τους αναζητούντες άσυλο. Αλλά οι αρχές των Ηνωμένων Εθνών, μάλλον ο εκπρόσωπος, ο απεσταλμένος, έπρεπε να φύγει από τη Λιβύη. Δηλαδή εκδιώχθηκε ο ύπατος αρμοστής από τη Λιβύη σε σχέση με το θέμα των αναζητούντων άσυλο. Πώς ε, εξελίσσεται αυτή η κατάσταση που είναι άκρος ανησυχητική, δηλαδή το ότι εκδιώχθηκε ο ε, ύπατος αρμοστής από τη χώρα που μπορούσε να ελέγξει κάπως την κατάσταση σε σχέση με τους ε, μετανάστες. Και ποια άλλη λύση συμβιβασμού βλέπετε. Για τη μετανάστευση θα υπάρξουν και άλλα ερωτήματα και θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω κατά πόσο διαβάσατε την ε, τελευταία έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για τη Λιβύη, η οποία εκδόθηκε αυτές τις ημέρες. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να διαβάσω πλήρως το κείμενο. Γίνεται μνήα και σε αυτό το θέμα των ετούντων άσυλο και των μεταναστών και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ιδιαίτερα για την εξέλιξη αυτού του ζητήματος. Ως προς το κεφάλαιο για το εμπόριο, όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και μας είπατε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Λιβύη είναι εκτός του συστήματος του ΠΟΕ και δεν κατανοεί τους κανόνες λειτουργίας αυτού του πλαισίου. Είπατε ότι υπάρχει θέληση εξοικείωσης με αυτό το σύστημα, αλλά έμπρακτα υπάρχουν δυσκολίες και ασυνενοησία σε σχέση με το standstill clause. Αυτές είναι οι ερωτήσεις αυτή τη στιγμή. Πρέντα για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με πολύ γενναιόδωρος χρόνο στα τρία λεπτά δεν το ήλπιζα καν. Ευχαριστούμε κύριε Μιγκαρέλη για την περιγραφή σας των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να επιμείνω σε ένα σημείο διότι την προηγούμενη εβδομάδα όπως θα ξέρετε στο Στρασβούργο δεχτήκαμε ένα ψήφισμα για το λεπτό θέμα των εκτελέσεων στη Λιβύη. Είχαμε πληροφορίες που μάθαμε και από τον τύπο στη Λιβύη που επιβεβαιώνουν την εκτέλεση τουλάχιστον 18 ατόμων μεταξύ των οποίων και ξένων. Και οι οποίοι δεν έτυχαν της θεούσας νομικής προστασίας ή καμίας προστασίας. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εάν το θέμα της θανατικής ποινή συζητιέται και αυτό μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί όταν λέτε ότι υπάρχει πρόοδος για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ήθελα να ρωτήσω, συμφωνούν να υπάρξουν αλλαγές για εκδημοκρατισμό, γιατί για αυτούς δημοκρατία εννοεί τζαμαχηρία, όχι δυτική δημοκρατία. Όταν μιλάτε λοιπόν για ανθρώπινα δικαιώματα, συζητάτε και το θέμα της θανατικής ποινή, διότι η Λιβύη είναι γνωστό ότι έχει αρνηθεί να συνυπογράψει το ψήφισμα του ΟΗΕ κατά της θανατικής ποινής. Πράγμα βέβαια το οποίο συνδέεται και με τη μετανάστευση. Διότι μεταξύ των εκτελεστέντων το Μάιο λένε ότι υπήρχαν και πολίτες του Τσάντ, της Νιγηρίας και από Το καθεστώς του Καντάφη έχει καλές σχέσεις με τη Χούντα του Νίγηρα με το λοχαγό εκεί που είναι επικεφαλής και υπάρχουν και πολίτες του Τσάντ και άλλοι όπως είπα που εκτελέστηκαν και που διατρέχουν μεγάλους κινδύνους από τις αρχές της Λιβύης. Απλό το ερώτημα λοιπόν. Η θανατική ποινή και το καθεστώς των αλλοδαπών συζητιούνται και αυτά μεταξύ των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε κύριε Πρέντα. Σεβαστήκατε και το χρόνο σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λόκμπιλερ. Κυρία, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ και εγώ στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσείς κύριε Μινγκαρέλη, είπατε ότι έχετε σημειώσει και επιτυχίες. Σας συγχαίρω γι' αυτό. Είπατε ταυτόχρονα ότι η στάνταρντ ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα έγινε μεν δεκτή, αλλά το ζήτημα είναι πώς θα εφαρμοστεί και αν θα εφαρμοστεί στην Λιβύη. Εν προκειμένου είπατε ότι η Λιβύη εξακολουθεί να μην θέλει να κυρώσει τη συνθήκη της Γενέβης, από την άλλη μεριά έχει δεχτεί να μην εκδίδει μη ε, Λιβύους πρόσφυγες. Έχουμε όμως πληροφορίες ότι υφίστανται βαριές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους. Επίσης, όπως είπε και η κυρία Γκόμες, φαίνεται να υπάρχει ένα ταμπού της λιβικής κυβέρνησης σχετικά με το ενδεχόμενο κύρωσης του καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου. Στην Καμπάλα προμηνώς κάναμε μια σχετική διάσκεψη. Υπάρχει ένας νέος ορισμός, ασθενής μεν, αλλά νέος, σχετικά με τον επιθετικό πόλεμο. Και εφόσον δηλαδή αρχίζει κανείς ένα επιθετικό πόλεμο, θεωρείται αυτό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και επομένως εμπίπτει στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου αυτού. Τώρα υπάρχουν και άλλες κυβερνήσεις στην Αφρική που έχουν και διαφορετική θέση. Ποια είναι η θέση της ε, λιβικής κυβέρνησης εν προκειμένου. Σας ευχαριστούμε για Λόχ Μπίλερ. Μίλαν μόνο. Σας ευχαριστώ κύριε Μιγκαρέλη που ξαναήρθατε στο Κοινοβούλιο για άλλη μια φορά. Θα ήθελα καταρχήν να μας μιλήσετε για το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας, διότι νομίζω ότι έχει επιτελεστεί μεγάλη πρόοδος. Για τη Λιβύη υπάρχει μία κόκκινη γραμμή σε σχέση με τους μετανάστες που προέρχονται από τρίτες χώρες. Αυτό θα ήταν ένα πολύ κακό προηγούμενο για τις διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο. Και δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να γίνει επανεισδοχή των παρανόμων μόνο για την περίπτωση της ε, Λιβύης. Ε, δεν υπάρχει ε, μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού όπως υπάρχει στην, στο Μαρόκο και στην Αλγερία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι κάνει αυτή τη στιγμή η Λιβύη με τους ε, μετανάστες που προέρχονται από τρίτες χώρες και μεταβαίνουν στην Ιταλία, διότι επί του παρόντος πρέπει να το επιλύσουν οι Ιταλοί το θέμα από ό,τι φαίνεται. Επίσης, ποια είναι η στάση σε σχέση με την Ένωση για τη Μεσόγειο. Υπάρχει μία ε, αμφιθυμία θα μπορούσα να πω ως προς τη διαδικασία της ε, Βαρκελόνης από τους ε, Λιβύους, από τους Λίβιους. Σε σχέση με το κεφάλαιο της ενέργειας θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με μία ε, πρόταση πλαίσια. Από όσο γνωρίζω, η, Ισπανική Προεδρία θα μεταβεί στη Λιβύη αύριο μέσα στα πλαίσια μιας ενδεχόμενη διμερού συμφωνίας. Γνωρίζετε κάτι επί του θέματος. Ευχαριστούμε κύριε Μίλαν Μον. Πριν συνεχίσουμε με τη συζήτηση, θα ήθελα να καλωσορίσω εξ ονόματος ημών μίας αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου της Ινδονησίας υπό τον Κεμάλα Ζη Ταμποέλ που είναι πρόεδρος της ε, πρώτης επιτροπής βρίσκονται εδώ στις Βρυξέλλες στα πλαίσια μιας διακοινοβουλευτικής συνάντησης με το κοινοβούλιο μας. Ελπίζω η συνάντηση αυτή να είναι ιδιαίτερα παραγωγική και να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες εξελίξεις στις σχέσεις μας για μια γενικότερη αμοιβαία κατανόηση. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει μία συμφωνία εταιρικής οικονομικής σχέσης που υπεγράφει το 2009 με την Ινδονησία και με αυτή σας την παρουσία ελπίζω να φτάσουμε σε θετικές εξελίξεις για όλους. Ο κύριος Κυρίλοφ έχει το λόγο για τρία λεπτά. Grazie, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την πλήρη ενημέρωση που μας έδωσε ο κ. Μινγκαρέλη. Δεν έχω ιδιαίτερες ερωτήσεις γιατί για μένα τα πράγματα είναι αρκετά σαφή. Το εμπόριο όχι. Διεθνές ποινικό δικαστήριο όχι. Έκδοση ε, αλλοδαπών παράνομων μεταναστών, όχι. Και μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό και ως μοχλός. Εάν δεν συμφωνηθεί, μπορεί κατά κάποιο τρόπο να είναι ένα εργαλείο που θα έχουν στα χέρια τους για να μας εκβιάσουν. Πριν να μιλήσουμε όμως για ανθρώπινα δικαιώματα, να πω το εξή. Εν τέλει, ποιο είναι το ενδιαφέρον μας, ποιοι είναι οι στόχοι μας για την συμφωνία αυτή. Έχετε μέχρι τώρα, όπως είπατε, επτά γύρους διαπραγματεύσεων. Μπράβο, αλλά τι πετύχατε. Δεν σας μέμφωμαι ούτε εσάς ούτε την Κομισιόν. Γνωρίζω καλά πόσο αδίστακτο είναι αυτό το καθεστώς στην περίπτωση των νοσοκόμων από την Βουλγαρία που κρατήθηκαν εκεί επί χρόνια που αντιμετώπιζαν την ποινή του θανάτου επειδή υποτίθεται ότι σκότωσαν παιδιά στα νοσοκομεία. Και ευτυχώς τέλος πάντων γλίτωσαν, επέστρεψαν στη Βουλγαρία μετά από την επίδειξη αυτή ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Τα ίδια πράγματα επαναλαμβάνονται τώρα με Ελβετούς υπηκόους είναι κατά κάποιο τρόπο όμοιροι. Ξε, ξεχάστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξεχάστε τις δίκες, δίκες. Λυπούμε πολύ που η χώρα τόσο απεισιόδοξα, αλλά δεν υπάρχει άλλη χώρα με τέτοιο αδίστακτο καθεστώς όπου ε, στην πραγματικότητα συνδυάζει την δημαγωγία και την δικτατορία με τόσο επιτυχημένο τρόπο θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ξεκαθαρίσουμε ποιοι στόχοι, ποιοι είναι οι στόχοι μας. Εγώ δεν ξέρω άλλη χώρα, άλλο καθεστώς το οποίο να συλλαμβάνει αλλοδαπούς υπηκόους, να τους κρατάει ομήρους και επίσης να μοιράζει τόσο απλόχερα τις θανατικές καταδίκες. Ευχαριστώ κύριε Κυριλόφ. Άτκινς, τρία λεπτά. Πρόεδρε, εγώ είμαι υπέρ της σύναψης αυτής της συμφωνίας. Ξέρουμε ότι η Λιβύη έχει τα προβλήματά της και δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στις δικές μας προσδοκίες, αλλά γνωρίζοντας την ιστορία θα ξέρετε ότι η Λέπτης Μάγνα έχει παίξει μαζί με άλλες αρχές πόλεις πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τη συμφωνία αυτή. Έχω όμως και εγώ ένα ερώτημα. Η Βρετανία όπως και πολλές άλλες χώρες είχε προβλήματα με τρομοκράτες που μάλλον προέρχονταν από τη Λιβύη. Τώρα θέλουν να συμμετάσχουν στη ζωή της διεθνούς κοινότητας. Είστε πλήρως ικανοποιημένοι ότι οι δεσμεύσεις τους κατά της τρομοκρατίας είναι ειλικρινείς και αποδεδειγμένες και ότι τώρα θα μπορέσουν να γίνουν σύμμαχοι αντί εχθροί. Ευχαριστούμε κύριε Άτκινς. Θα δώσω το λόγο τώρα στον δόκτωρα Μιγκαρέλη για πέντε λεπτά αν είναι δυνατόν για να απαντήσει και μετά θα περάσουμε στη δεύτερη φάση της συζήτησης. Παρακαλώ όλοι να σεβαστούν το χρόνο τους. Ορίστε δόκτωρα. Ευχαριστώ. Αρχίζω με την ερώτηση κυρίας Γκομές. Για τα νομικά πρέπει να σας πω όπως μου όπως πρέπει να το κάνω ότι οι υπηρεσίες της Κομισιόν θα προτείνουν τη νομική βάση στο τέλος της διαπραγμάτευσης όταν θα ξέρουμε ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας. Όταν θα γνωρίζουμε δηλαδή τι τύπος συμφωνίας είναι θα καθορίσουμε και τη νομική της βάση. Μπορώ απλώς να σας πω ότι δεν πρόκειται καθόλου για προσπάθεια μείωσης του ρόλου του Κοινοβουλίου Έχω έρθει πολλές φορές να σας πληροφορήσω, σας λέω καθαρά ποια είναι τα προβλήματα. Λαμβάνουμε υπόψη τις δηλώσεις, προτάσεις και σχόλιά σας, αλλά επαναλαμβάνω ότι οι νομομαθείς θα το καθορίσουν και εγώ δεν μπορώ να τα αλλάξω. Για το καθεστώς της Ρώμης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Στόχος μας είναι, επαναλαμβάνω, όλες οι χώρες με τις οποίες έχουμε εταιρική συμφωνία να δεχτούν, να συμμετάσχουν στη λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και στο καθεστώς της Ρώμης. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Πάρα πολλές χώρες εταίροι μας και πολλές σημαντικές και στρατηγικές δεν συνεργάζονται, δεν είναι τμήμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Δεν το θέλουν ούτε και οι Λίβοι, αλλά δεν είναι οι μόνοι. Έχω διαπραγματευτεί συμφωνίε και με άλλες χώρες που τις θεωρούμε πολύ καλούς εταίρους και δεν θέλουν ούτε να τα ακούσουν. Δεν είναι λοιπόν λόγος να, να πάψουν οι διαπραγματεύσεις Μην το θεωρήσετε λοιπόν ιδιαιτερότητα της Λιβύης, δεν θα ήταν ε, αληθές αυτό. Όταν είπα ότι υπάρχει πρόοδος, το γεγονός, εννοούσα ότι το γεγονός και μόνο ότι οι Λίβοι δέχονται μια παραπομπή όπου να λένε ότι αναλαμβάνουν τη δέσμευση μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταπολεμήσουν τα σοβαρότερα, τα ιδεχθέστερα εγκλήματα όπως εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίες είναι είπα ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση δεν θα πει ότι είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι εξάλλου η εντολή μας δεν είναι να είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι αλλά δεν μας είπαν και ότι το αποκλείουν είπαν λοιπόν, θα το συζητήσουμε δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι αλλά δέχτηκαν να κάνουν ένα βηματάκι. Επίσης τώρα για τους αιτητές ασύλου και τους πρόσφυγες δεν έχουν καμία πρόθεση να δεχτούν τη συμφωνία της Γενέβης του 51 αλλά, τη συνθήκη της Γενέβης, αλλά δέχονται να γίνει παραπομπή στην αναγκαιότητα να διασφαλιστεί μια προστασία των μεταναστών που χρήζουν διεθνούς προστασίας λέει. Και πάλι δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Θα θέλαμε κάτι πολύ περισσότερο, αλλά αυτό πετύχαμε μέχρι τώρα. Δεν μας έδωσαν αυτό που θέλαμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι όπως λέτε κύριε Κυρίλοφ δεν μας έδωσαν nothing. Δεν είναι αλήθεια. Για την υπάτη αρμοστία. Έκλεισαν την αντιπροσωπεία εκεί. Πήγαμε επιτόπου μετά από μερικές μέρες και τους είπαμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο, ιδίως σε μια χώρα όπου υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες και αιτητές ασύλου και μας εξήγησαν ότι η αντιπροσωπεία αυτή βρισκόταν σε νομικός άτυπον καθεστώς. ότι δηλαδή δεν είχαν κάνει αυτά που έπρεπε για να ζητήσουν νομικό καθεστώς αναγνωρισμένο και πολλοί μας είπαν ότι η αλήθεια ήταν αυτό. Για μας βέβαια παραμένει απαράδεκτο να κλείνουν την αντιπροσωπεία της ΥΠΑ της Αρμοστίας και τους είπαμε με διάφορους τρόπους τη θέση μας αυτή. Υπάρχει μια αντιπροσωπεία της έδρας του ΟΗΕ στη Γενέβη που θα πάει στη Λιβύη και θα προσπαθήσει να τα τακτοποιήσει όλα αυτά, να δεχτούν οι Λίβοι, δηλαδή να ξανανοίξει το γραφείο της αντιπροσωπείας της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Δεν ξέρω αν θα λήξουν θετικά αυτά, αλλά το είπαμε, το συζητήσαμε και τους ζητήσαμε να το συζητήσουν με την αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ. Την έκθεση της αμνηστίας όχι δεν την διάβασα, ευχαριστώ για την πληροφορία, θα το διαβάσω. Για τα εμπορικά προβλήματα όπως σας είπα υπάρχει το ότι δεν δέχονται το πάγωμα των δασμών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ούτε είναι βέβαιο ότι θα δεχτούν τις βασικές αρχές του ΠΟΕ στο τελικό κείμενο της συμφωνίας. Ακριβέστερα μου λένε οι συνάδελφοί μου ότι υπάρχουν προβλήματα επίσης και για τις δημόσιες αγορές, ότι για τις υπηρεσίες δεν υπάρχει εθνική στρατηγική καμία και γι' αυτό είναι δύσκολο να πούμε ότι θα δεχτούν δεσμεύσεις. Για την ενέργεια υπάρχουν δυσκολίες και για τις συναλλαγές δεν υπάρχει καμία καθορισμένη και σαφής δασμολογική πολιτική. Δεν υπάρχει καμία βάση διαπραγμάτευσης λοιπόν. Κύριε Πρέντα τώρα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τις εκτελέσεις και εμείς καταδικάσαμε τις εκτελέσεις αυτές. Στην Τρίπολη η Ισπανική Προεδρία έκανε ένα διάβημα, αλλά στα πλαίσια της συμφωνίας τίποτα δεν αναφέρεται ούτε στην κατάργηση της θανατικής ποινή, ούτε στο πάγωμά της ή μορατόριουμ αλλά το ίδιο ισχύει για όλες τις εμπορικές μας συμφωνίες δεν γίνεται λόγος για τέτοια στα πλαίσια όμως του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές που δέχτηκαν οι Λίβοι κάθε φορά τους μιλάμε για την αναγκαιότητα να καταργηθεί η θανατική ποινή ή τουλάχιστον αμέσως να εφαρμοστεί μορατόριο όπως γίνεται και με τις άλλες χώρες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μεταχείριση των προσφύγων στη Λιβύη δεν είναι καλή αυτή η μεταχείριση προφανώς. Αλλά στόχος μας δεν είναι να λύσουμε το πρόβλημα των δυστυχισμένων αυτών ανθρώπων αλλά να δημιουργήσουμε μια βάση που να επιτρέπει τον τακτικό διάλογο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λύσουμε τις διαφορές μας αν δεν συζητάμε. Με καταδίκες δεν γίνεται τίποτα. Μόνο με τακτικές συζητήσεις. Αρκούν οι συζητήσεις όχι, αλλά σε μια συζήτηση μπορεί κανείς τουλάχιστον να μιλήσει για μια στρατηγική, να τους πούμε αν θέλετε κάτι που σας ενδιαφέρει, όπως ας πούμε συνεργασία για ορισμένους τομείς διαχείρισης των μεταναστών, τότε και εσείς πρέπει να κάνετε ορισμένες υποχωρήσεις. Αν δεν υπάρξει τέτοια συζήτηση και διαπραγματεύση που προς στιγμή δεν υπάρχει, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Δεν σας λέω λοιπόν ότι το, η ύπαρξη μια συμφωνία θα λύνει τα προβλήματα καθεαυτή. Να. Αλλά δίνει μια παραπάνω ευκαιρία την οποία τώρα δεν έχουμε. Για το καθεστώς της Ρώμης. Μα σας το είπα. Κι άλλοι εταίροι μας δεν το δέχονται. Δεν πάβουμε να τους το ζητάμε, αλλά δεν είναι πάλι λιβική ιδιαιτερότης. Καμία χώρα δεν δέχεται τις επανεισδοχές των μεταναστών όπως ζητάτε. Με τη Ρωσία και την Ουκρανία το πετύχαμε, αλλά πρώτα με μεταβατικές περιόδους 2-3 ετών και έπειτα είχαν ως αντίτιμο και μία διευκόλυνση του καθεστώτος των θεωρήσεων η επίσκεψη της Ισπανικής Προεδρίας κατά εμάς ήταν διμερές θέμα. Συζήτησαν και για το πρόβλημα με τους Ελβετούς. Δεν λύθηκε το πρόβλημα αλλά το συζήτησαν. Ο στόχος το έχω πει ποιο είναι, να δημιουργηθεί η βάση ενός διαλόγου μας δίνει μια ευκαιρία προόδου. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση βέβαια. Αν όμως θέλουμε να υπάρξει ευκαιρία πρέπει να συνομιλούμε. Αν δεν συνομιλούμε δεν λύνουμε τίποτα για την καταπολέμηση της τυρομοκρατίας. Δεν έχω καμιά πληροφορία που να μου επιτρέπει να πω ότι κάνουν ό,τι πρέπει για να την καταπολεμήσουν, αλλά μπορώ να σας πω ότι κατά τις συζητήσεις μας πάντοτε επιμένουν ότι είναι αποφασισμένοι να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές της τρομοκρατίας και ιδίως να εφαρμόσουν με μας συνεργασία συγκεκριμένη για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία τουλάχιστον στο τμήμα της Βορείου Αφρικής και της υποσαχαρίας τη αυτής για καταπολέμηση της τρομοκρατίας εκεί. Άρα από την πλευρά των δεσμεύσεων υπάρχουν δεσμεύσεις αλλά δεν μπορώ να σας πω αν επί που τα εφαρμόζουν όλα αυτά δεν έχω στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, δόκτωρα Μιγκαρέλη. Δυστυχώς για το δεύτερο μέρος των συζητήσεων, επειδή πρέπει να κλείσουμε μέχρι τις 11, θα πρέπει να σας ε, διακόψω, και, μάλλον να σας δίνω το λόγο για 1,5 λεπτό και όχι 3 ε, λεπτά. Χαίρομαι που το ανακοινώνετε όταν λαμβάνω εγώ το λόγο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κύριε Μιγκαρέλη, εκπλήσωμε που σας ακούω γιατί για το γραφείο του ΙΠΑ του Αρμαστού το ακούμε από εσά ε, ότι ποτέ δεν ε, έκανε, μάλλον ποτέ δεν ζητήθηκε ε, επίσημη άδεια εγκατάστασης. Εγώ ξέρω ότι αυτό μας λένε οι Λίβοι εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν ισχύει. Όταν απευθύνεστε σε βουλευτές, να λαμβάνετε υπόψη την κατάσταση όπως πραγματικά ισχύει. Δηλαδή να μας πείτε γιατί εκδιώχθηκε ο ύπατος αρμοστής από τη Λιβύη και να έρθετε σε επαφή και με το γραφείο της ύπατης Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών εδώ. Βεβαίως υπάρχουν πολλές χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε στενά που παραβιάζουν ε, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση της Ρώμης. Αλλά μέσα στα πλαίσια των ακροβασιών αυτών των διαπραγματεύσεων και είμαι σίγουρη ότι κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Αν όμως φτάσουμε σε μία ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή μία ε, ρήτρα που δεν φτάνει στη σύμβαση της Ρώμης, αλλά που αναγνωρίζει τις γενοκτονίες. Κύριε Πρόεδρε, δεν κάνετε τίποτα γιατί εσείς παραβιάζετε το διεθνές δίκαιο όπως την αρχή της μη ε, εκδίωξης. Δεν σας δίνω, δεν δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερο χρόνο. Βερτζάτ, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, είμαι η πρώτη ομιλήτρια από την ομάδα μου και γι' αυτό θα ήθελα τουλάχιστον ένα λεπτό. 1,5 λεπτό, ορίστε. Ναι, αλλά είναι σκανδαλώδες να μην αφήνετε πρώτα να λάβει το λόγο τουλάχιστον ένας ομιλητής από κάθε ομάδα. Έτσι κάνουμε συνήθως. Και μη μετρήσετε το χρόνο μέχρι τώρα, παρακαλώ. Λοιπόν, μας μιλήσατε για προόδους και για αδιαπραγμάτευτα θέματα για τους Λίβιους, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Συνθήκη της Γενέβης. Απ' την άλλη μεριά ακούμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία αν δεν δεχτούν τη Συνθήκη της Γενέβης. Τώρα μα λέτε ότι αλλάζει αυτό, ότι δεν θα είναι εμπόδιο. Όσοι δεν δέχονται να προσαχθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μεταξύ των οποίων και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί δεν πρέπει να υπογράφουν τέτοιες συμφωνίες μαζί μας. Για την υπάτη αρμοστία η Ελένη Φλότρα μας είπε ακριβώς τι ισχύει, ας μην επανέλθω λοιπόν. Με όλο το σεβασμό λοιπόν που ο φίλος εκπρόσωπο της Κομισιόν αναρωτιέμαι αν είστε αφελείς, αν το κάνετε επίτηδες ή αν μας κοροϊδεύετε. Διάβασα την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Οι διαπραγματεύσεις έχουν κρατήσει μήνες με τη Λιβύη. Υπάρχουν κι άλλες εκθέσεις από αυτό. αν δεν διαβάζετε τις εκθέσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων, διαβάστε το διεθνή τύπο που μας γελιοποιεί παντού. Πώς μπορείτε να πιστεύετε ότι είναι δυνατόν με τον κύριο Καντάφη να υπάρξει πρόοδος. Συνομιλείτε με αυτόν τον δικτάτορα σαν να ήταν δημοκράτης, ενώ δεν είναι. Ρωτήστε τους Ελβετούς και θα μάθετε τι διάλογος υπάρχει με τη Λιβύη. Και αυτοί υποχώρησαν σε όλα. Ο κύριος Μπεναράμπα του. Η κυρία. Η κυρία. Οι συνάδελφοι υπέβαλαν πολλές ερωτήσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τη Σύμβαση της Γενέβης. Δεν θα επανέλθω επ' αυτού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως κατά πόσο θα μιλήσετε, θα διαπραγματευτείτε την κατάσταση των γυναικών και έχετε εγγύσεις ως προς τα δικαιώματα των γυναικών και της οικογένειας γενικότερα. Το δεύτερο μου ερώτημα αφορά τη γεωγραφική θέση της Λιβύης που βρίσκεται στο Μαγκρέμπ. Λάβατε υπόψη αυτή την ε, θέση της Λιβύης, Λιβύης που κατέχει μέσα στα πλαίσια της περιφέρειας του ε, Μαγκρέμπ. Ο κύριος Παντζέρη για 1,5 λεπτό. Δεν έχω καμία αμφιβολία ως προς τις ε, δυνατότητες διαπραγμάτευσης της Επιτροπής. Έχουν γίνει θετικά βήματα αλλά δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι μπορούμε να συμμεριστούμε απόλυτα την αισιοδοξία σας, κύριε Μιγκαρέλη. Μας ενδιαφέρουν βεβαίως και οι δυνατότητες μιας διμερούς συμφωνίας σε, στον τομέα του εμπορίου, οικονομικών ζητημάτων και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να συνάψουμε μια συμφωνία διότι αυτό θα μας βοηθήσει, αλλά δεν είναι κάτι το υποχρεωτικό. Τρεις είναι οι ερωτήσεις. Όταν μιλάμε για διμερείς ε, συμφωνίες μεταξύ κρατών, συνεισφέρουν ή αποτελούν τροχοπέδι στις διαπραγματεύσεις. Διαφορετικά θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη αυτά να σταματήσουν τις διαπραγματεύσεις μέχρι ότου καταφέρουμε και φτάσουμε σε μια Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Ως προς το θέμα της επανεισδοχής, θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο ε, πρόβλημα σε σχέση με αυτό το σκέλος της συμφωνίας. Σας γνωρίζω πολύ καλά, αλλά από πλευράς ε, Κοινοβουλίου χρειαζόμαστε κάποια τεκμηρίωση που να μας δείχνει πώς προχωρούν αυτές οι διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να έχουμε κάτι γραπτός και να μην αρκεστούμε στις ακροάσεις. Ε, έχει λήξει ο χρόνος ε, για τη συζήτηση αυτή, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να απαντήσετε. Ιδιαίτερα μετά από ε, ορισμένα ιδιαίτερα δεικτικά σχόλια που έγιναν. Ως προς την κυρία Φλότ, σε σχέση με την Λιβύη και τη θέση της απέναντι στον ΙΠΑ το αρμοστή, είπα ότι ε, οπωσδήποτε αντιταχθήκαμε στο κλείσιμο του, του γραφείου της ΙΠΑ της αρμοστίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είπα ότι κάτι τέτοιο δικαιολογείται. Είπα ότι θα πρέπει να ανοίξει το ταχύτερο δυνατόν και ζητήσαμε να ε, μεταβεί αντιπροσωπεία από τη ε, Γενέβη στη Λιβύη για να επαναδιαπραγματευτεί το θέμα. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα να σας πω ναι είναι απαράδεκτο χωρίς να σας πω ποια είναι και η αντίθετη γνώμη. Αν θέλετε αυτό θα κάνω την επόμενη φορά. Ως προς την ενδιάμεση ρήτρα προς που οδηγεί στην κατάρριψη του διεθνούς δικαίου, θα το αναφέρουμε στα πλαίσια της εντολής μας. Είναι ένα πραγματικό ζήτημα. Κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις διεθνείς ρήτρε όπως προϋπάρχουν ή θα πρέπει να προσπαθήσουμε από καιρού εις καιρών, ακόμα και αν δεν λαμβάνουμε αυτό που θέλουμε, μία ενδιάμεση ρήτρα. Αυτό είναι ένα θέμα ουσίας. Κυρία Βερζά, αν είμαι αφελής ε, ε, ή αν σας ε, κοροϊδεύω, σίγουρα δεν σας κοροϊδεύω και διαλέξτε κατά πόσο είμαι αφελής ή προσποιούμε ότι είμαι αφελής. Ως προς τα δικαιώματα των γυναικών, βεβαίως το συζητήσαμε. Συζητήσαμε το θέμα και με γυναίκες και θα ήθελα να σας πω ότι το καθεστώς έναντι των γυναικών είναι πολύ πιο προστατευτικό έναντι άλλων χωρών και θα υπάρξει μια ειδική μνήα για την διάθεση βελτίωσης της κατάστασης των γυναικών, των δικαιωμάτων των παιδιών σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό που επιθυμούμε, το συζητούμε όμως γιατί δεν δέχονται το σημείο εκκίνησης, το δικό μας δηλαδή, ότι η κατάσταση των γυναικών στη Λιβύη δεν είναι μια κατάσταση που γίνεται αποδεκτή από εμάς. Για τον κύριο Παντζέρη, διμερείς συμφωνίες, τροχοπέδι ή όχι, ναι, συχνά πρόκειται για ένα μεγάλο πρόσχομα, διότι όταν μιλάμε για τις μεταναστευτικές ροές, με την Λιβύη ή το Μαρόκο για θέματα θεωρήσεων ή επανεισδοχής, επειδή υπάρχουν διμερείς συμφωνίες με τους Ιταλούς, τους Γάλλους και τους Ισπανούς, για αυτούς διευθετείται το μεγαλύτερο μέρος του ζητήματος. Γι' αυτό είναι δύσκολο να φτάσουμε σε κοινοτικέ συμφωνίες. Επανεισδοχή. Δέχονται να ε, μπουν οι Λίβοι υπήκοοι που βρίσκονται παράνομα στο δικό μας έδαφος, όχι όμως τους υπηκόους τρίτων χωρών, δηλαδή έναν Νιγηριανό ή έναν ε, κάτοικο από την Μπουρκίνα Φάσο. Δεν θέλουν να μεταβούν αυτοί οι υπήκοοι να περάσουν από το δικό τους έδαφος. Και αυτό είναι ε, μια μεγάλη τροχοπέδη, διότι τους λέμε να δεχτούν όλους τους μετανάστες που βρίσκονται παράνομα στο ευρωπαϊκό έδαφος. Εάν θέλουμε να κερδίσουμε όμως θα πρέπει να διευρύνουμε το ζήτημα της μετανάστευσης με μια, υπό μια ευρύτερη έννοια λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα, ε, τις διάφορες συνιστώσεις του θέματος της ασφάλειας. Ως προς το τελευταίο ερώτημα, θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να σας στείλουμε ε, κείμενα. Πρέπει να το συζητήσω με το Συμβούλιο. Αλλά θα το λάβω σοβαρά υπόψη. Ωραία. Ευχαριστούμε τον δόκτωρα Μιγκαρέλη. Πολύ καρποφόρα αυτή η συζήτηση. Και θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να ξαναξετάσουμε το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Και περνάμε στο δεύτερο σημείο. Ο δόκτωρ Μορέλ, ειδικό απεσταλμένος Ευρωπαϊκής, ειδικός εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία, θα ήθελα να έρθει εδώ στα, στα έδρανα της Προεδρίας. Τον περιμένουμε. Qualche minuto per farlo arrivare. Ο κύριος Μορέλ είναι μαζί μας. Αρχίζουμε με τη συζήτησή μας ως προς την κατάσταση στο Κυργιστάν με τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Κεντρικής Ασίας αυτή η συνάντηση είναι αναγκαία. Αν και βρισκόμαστε συχνά με τον δόκτορα Μορέλ, όμως γνωρίσαμε μία πρωτόγνωρη βία στο Κυργιστάν πρόσφατα, στις 10 Ιουνίου. Στην πόλη Ως μιλάμε για 191 νεκρούς, για 1.900 τραυματίες και ίσως ο αριθμός να είναι πολύ υψηλότερος από τον ε, παραδεχόμενο και υπάρχουν και πολλοί πρόσφυγες προς το Ουσμπεκιστάν. Μιλάμε για 500.000 ε, πρόσφυγες προς το Ουσμπεκιστάν. Έχουμε εγγράψει 5 εκατομμύρια ευρώ για επίγουσα βοήθεια. Στις 11 Ιουνίου η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, η ύπατη εκπρόσωπος, η κυρία Άστον, προέβησε μία δήλωση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου ε, προέβαλε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την προσωρινή κυβέρνηση για την αποκατάσταση της νομιμότητας και ενθάρρυνε τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να σταθεροποιηθεί πολιτικά η κατάσταση στη χώρα. Ελπίζουμε και το δημοψήφισμα που βλέπετε για τις 27 Ιουνίου για το ε, Σύνταγμα να ε, σέσει ο πέρας και προβλέπονται και βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο, όπως γνωρίζετε. Στις 14 Ιουνίου, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών έγινε μια ειδική δήλωση επί του θέματος. Ο δόκτωρ Μορέλ έχει μεταβεί στο Κυργιστάν και μπορεί να μας δώσει μια ακριβή εικόνα της κατάστασης και θα μας μιλήσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Το θέμα είναι ευρύτατο, αλλά θα ήθελα να αρκεστείτε στα 10 λεπτά, έτσι ώστε μετά να γίνει συζήτηση. Σας δίνω το λόγο λοιπόν και θα σας ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρονικό όριο που μου επιβάλλεται. Γνωρίζω και πόσο αυστηρό είστε και βεβαίω έχω ενδιαφέρον να προβούμε μετά σε ανταλλαγή απόψεων. διεξάγεται αυτή τη στιγμή συνεδρίαση του ΚΟΠΣ. Θα δούμε βέβαια μετά ότι πρέπει να πάω ε, να ε, συμμετάσχω σε αυτή τη διάσκεψη που διεξάγεται ταυτόχρονα. Πρόκειται για ένα θέμα ε, βαρύτατης σημασίας διότι εκτός από την μοίρα της χώρας αυτής ε, θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα ολόκληρη της περιοχής αυτής της Κεντρικής Ασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμμετάσχει πιο μεθοδικά και πιο δραστήρια εδώ και 3,5 χρόνια περίπου αναπτύσσοντας μια στρατηγική για την Κεντρική Ασία με στόχο μια πιο μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση. Βρισκόμαστε λοιπόν απέναντι σε μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση και πρέπει να παίξουμε ένα ρόλο ενός φορέα που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην σταθεροποίηση της περιοχής. Έχουμε δημιουργήσει ε, σιγά σιγά βήμα βήμα μια ε, εταιρική σχέση και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά σε μια τόσο σοβαρή κατάσταση. Τι συνέβη ακριβώς. Θα προσπαθήσω να ε, δώσω μια αρχή ανάλυσης της κατάστασης αυτής. Για να κατανοήσουμε την κατάσταση απέναντι στην οποία βρισκόμαστε, πρέπει να κατανοήσουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια κρίση η οποία πέρασε από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν η αλλαγή της εξουσίας στην Μπισκέκ μετά από τα γεγονότα που ούτως ή άλλως ήταν δραματικά με πάνω από 80 νεκρούς στο Μπισκέκ στις 7 Απριλίου. Πρόκειται για μια καμπή την οποία δεν ε, περιμέναμε οι περισσότεροι ευνηδιάστηκαν και η οποία έβαλε τέλος σε μια προεδρία την οποία ήταν μια υπόθεση ε, ε, ενός κλάν, μιας οικογένειας εν πάση περιπτώσει, του Μπακίερ που έγινε βέβαια η αλλαγή αυτή μέσα σε τραγικές συνθήκες έγινε μια πρώτη αλλαγή που ήταν ε, η επανάσταση της Τουλίπας η οποία τελικά δεν ε, ολοκληρώθηκε με τον πρόεδρο Ακαγεύ μπροστά σε αυτή την επιδείνωση της κατάστασης ε, διαρωτάται κανείς αν υπάρχει ίσως ένας κύκλος που ξεκινά από κάποιες ε, ελπίδες, και προσδοκίες του κόσμου, περνά από μια φάση μετά εναλλαγής κάποιων δυνάμεων που είναι μάλλον λίγο πολύ σταθερές με ένα ε, κομματικό πεδίο ευρύτατο και μετά η σώρευση κινημάτων από κάθε κατεύθυνση να δημοκρατία λένε καμιά φορά στην, ε, στα ρωσικά που είναι δημοκρατία των δρόμων με ταυτόχρονα κατάσχεση εντό εισαγωγικών της ε, εξουσία από μια προεδρία η οποία πάλι με την ε, ε, σειρά της προκαλεί κινήματα στους δρόμους και ξαναξεκινάει ο κύκλος αυτός. Βλέπετε δηλαδή μια κίνηση επαναλαμβανόμενη με ένα είδος χαρακτήρα μοιραίο. Η προσωρινή κυβέρνηση θέλει να ξεφύγει, να, να σπάσει αυτό τον φαύλο να ξεκινήσει ένα δημοκρατικό καθεστώς, αλλά αναγνωρίζει ίδια ότι πρέπει να αρχίσει από έκτακτες συνθήκες, η οποία αναστέλει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, λαμβάνει μέτρα επίγοντος χαρακτήρα. Εμείς ε, την ομάδα αυτή τη γνωρίζουμε αρκετά καλά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον διάλογό της με το Κυργιστάν και στην αποστολή που έχω αναλάβει εγώ ως ε, ειδικό εκπρόσωπος, ως ειδικό απεσταλμένος έχω έρθει σε επαφή τακτικά και με τις μη κρατικές οργανώσεις και με την ε, ε, αντιπολίτευση γενικά και μέσω της γερμανικής πρεσβείας έχουμε κατ' επανάληψη έρθει σε επαφή και με τα νέα μέλη και έχουμε υποστηρίξει την κυβέρνηση αυτή όταν αντιμετώπισε απειλές και φυσικές απειλές για να μπορέσουν να βγουν από τη χώρα. Έχουμε λοιπόν συνομιλητές οι οποίοι δέχονται ότι ναι μεν οι προσδοκίες τους είναι δημοκρατικές αλλά η κατάσταση είναι έκτακτη. Ταυτόχρονα υπήρξαν τάσεις στο Νότο γύρω από την ομάδα Μπακίεφ με πολλούς κινδύνους. Αυτό που κάναμε εκείνη τη στιγμή εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν να συνδιαλεχθούμε πολύ στενά και με τις άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται επί τόπου τον ΟΑΣΕ και τα Ηνωμένα Έθνη. Τρει επομένω ειδικοί απεσταλμένοι από την αρχή του Απριλίου σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου και τον Ιούνιο προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε για να αποφύγουμε τι επικαλύψεις, να περάσουμε τα ίδια μηνύματα και να επιτύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα επιτόπου. Το μήνυμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σαφέ. Είπαμε προτείναμε ένα οδικό χάρτη για την επιστροφή στη δημοκρατία ε, με κράτος δικαίου και με επιστροφή σε μια συνταγματική τάξη, πραγματικά δημοκρατική, μετά από αυτές τις ε, τραγικές εμπειρίες. Προσπαθήσαμε λοιπόν να μπούμε σε μια επαφή ε, προσεκτική με τις ε, επιτόπου αρχές, ο Καζαρμπαγεύ, πρωθυπουργός, δεν μπήκαμε στην παγίδα της αναγνώρισης γιατί δεν είναι αυτό το θέμα. Πρώτιστο μέλημα είναι η σταθεροποίηση. για να προωθήσουμε το Σύνταγμα αυτό για να αποφύγουμε να ξαναπέσουμε σε αυτή τη διαδοχή προεδριών που ξεκινούν όλες από, την ίδια, από το ίδιο κλάν με τήρηση των θεμελιωδών αρχών ενός κράτους δικαίου και αυτό είναι το κείμενο το οποίο θα υποβληθεί σε δημοψήφισμα την επόμενη Κυριακή. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθήσαμε να εργαστούμε μέχρι τη στιγμή που σημειώθηκε το δράμα της νύχτας της 10ης Ιουνίου όπου οδήγησε την κρίση σε μια δεύτερη φάση. Τι ακριβώς έγινε τη νύχτα της 10ης Ιουνίου. Ξεκίνησε μια σειρά επιθέσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ εθνο, εθνοτικών κοινοτήτων σε μια περιοχή του Νότου η οποία ήταν ήδη σε αναβρασμό αλλά μέχρι τότε είχε ε, κρατηθεί σε κάποια όρια με διάλογο μεταξύ των εκπροσώπων των εθνικών ομάδων. Όπως λέω, είχε συγκρατηθεί η αντίδραση αυτή, είχαν συγκρατηθεί αυτές ε, οι εκδηλώσεις βίας, ενώ ξαφνικά γενικεύθηκε η βία αυτή. Γιατί χωρίς αμφιβολία από έλλειψη επαγρύπνησης από πλευράς ε, της ΒΙΣΚΕΚ η έλλειψη αποτελεσματικότητας των δυνάμεων της ε, τάξης που αναγνωρίστηκε και από την προσωρινή κυβέρνηση και την κυρία Τουμπάγεβα που είναι η ε, προεδρεύουσα και της ομάδας Μπακίεφ που με κάποιο τρόπο συνέβαλαν. Υπενθυμίζω ότι ο πρόεδρος του πρόεδρου ε, Μπακίεφ έχει εγκατασταθεί τη γειτονική χώρα και από εκεί κινεί κάποια νήματα. Πρέπει να τεθεί το ερώτημα επίσης των δραστηριοτήτων εγκληματικών ομάδων, διότι το ή πολύ όσο αποτελεί ένα άξονα διακίνησης λαθεμπορίου ναρκωτικών έχουν γίνει προσπάθειες να αναλάβουν τα δίκτυα αυτά. Με, είναι, ε, υπάρχει αδυναμία των ε, κρατικών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Και αυτά είναι κάποια στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που δεν αποκλείονται. Ε, ο φανατισμός, ο ισλαμικός εξτρεμισμός, που είναι δυνάμεις που κυκλοφορούν στην περιοχή και έχουν διάφορα ονόματα τα οποία γνωρίζετε. Σήμερα ποια είναι τα ερωτήματα που τίθενται. Πρώτα, η συνέχιση της προσπάθειας νομοποίησης της κυβέρνησης και των θεσμών. Και αυτό είναι υπόθεση της ίδιας της κυβέρνησης του Κυρκιστάν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς για λογαριασμό τους. Εμείς εργαστήκαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο μαζί τους. Τώρα είναι οι επιλογές των τοπικών αρχών, των αρχών επιτόπου δηλαδή, και των ε, θεσμών του Κυργιστάν. Μετά η προσπάθεια να περάσουν σε εκλογές. Θα υπάρχουν παρατηρητές Υπάρχει επιτόπου ο πρέσβης Θερλέτς, ο οποίος ε, είναι επικεφαλής της διαρκούς αποστολής παρακολούθησης με ισχυρή παρουσία και του ΟΑΣΕ, με τη γνωστή του εμπειρία, και με υποστήριξη των αστυνομικών δυνάμεων για να αυξήσουν την ε, δυναμικότητά τους. Επίσης, το θέμα των συνόρων. Σημαντική κίνηση, όπως είπατε και εσείς, προσφύγων που πέρασαν στο Ουσμπεκιστάν, όπου ήταν αξιοσημείωτη η υποδοχή τους με οργάνωση γενικά πολύ καλή υποδοχή. κίνηση ήταν τέτοια, βέβαια, οι αριθμοί των προσφύγων ήταν τέτοιοι που ξεπέρασαν τις δυνατότητες υποδοχής του Ουσμπεκιστάν, το οποίο προσέφυγε σε διεθνείς οργανώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζητήσει την βοήθειά της και αναμένουμε τώρα η επιστροφή αυτών των προσφύγων οι οποίοι έφευγαν λόγω των απειλών αλλά και των πραγματικών επιθέσεων να δούμε τώρα πώς θα μπορέσουν να επιστρέψουν. Ήδη μιλούμε για μια επιστροφή 30-35.000 προσώπων. Αυτή είναι η πρώτη αριθμή, ενδεικτική αριθμή. Επίσης, το θέμα των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν, τη φαγή αυτή που διάρκεσε ορισμένε ημέρε, εδώ πρέπει να ρηχτεί άπλετο φως. Αυτή είναι και η επιθυμία της ίδιας της κυβέρνησης και βέβαια και η συμφιλίωση. Σε, όλη, σε όλη τη διάρκεια αυτών των τραγικών, των δραματικών ημερών υπήρχαν θαραλέοι Κυργίσοι οι οποίοι πήγαν να εργαστούν επί τόπου τον Ίκα για παράδειγμα και άλλα πρόσωπα που είναι σημαντικές μορφές της κοινωνίας των πολιτών ε, του Κυρκυζιστάν και που ήταν διαρκώς σε επαφή μαζί μας. Εν η διανομή βοήθειας. Υπάρχει επαρκής βοήθεια, αλλά πρέπει να φτάσει μέχρι τους απολύπτες που την χρειάζονται και να μπορέσουν έτσι να ξαναγυρίσουν στην καθημερινή ζωή τους. Έτσι θα αποφευθούν μελλοντικά προβλήματα. Θα πρέπει να νοικοδομηθούν τα σπίτια που καταστράφηκαν και ούτω καθεξής. Εν προκειμένου ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα ενός διαρκούς διαλόγου της υποστήριξης Τη προσπάθεια των αρχών για μια επιστροφή στη δημοκρατία. Επίσης, η ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη ανακοινώθηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ που προστίθεται στην βοήθεια που υπάρχει ήδη επιτόπου και που είναι τη τάξη των 6 εκατομμυρίων ευρώ στα πλαίσια του εργαλείου σταθερότητας με υποστήριξη πρωτοβουλειών της κοινωνίας των πολιτών και προγραμμάτων όπως αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Και τέλος, στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με τον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πέτερλε, που είναι εισηγητής για θέματα του Τατζικιστάν, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μορέλ για την ενημέρωση. Συμφωνώ με τη διαγνωσή σας. Εκφράζω βέβαια τη λύπη μου για το γεγονός ότι πέντε χρόνια μετά την πρώτη ανάληψη εξουσίας αντιμετωπίζουμε σήμερα μια πολύ δυσχερέστερη κατάσταση, μια πραγματική τραγωδία. Ο αριθμός των προσφύγων επίσης είναι πολύ υψηλός. Η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί εάν η διεθνής κοινότητα δεν δράσει με τρόπο αποφασιστικό. Συμφωνώ επίσης ότι είναι απαραίτητο να γίνουν δημοκρατικές αλλαγές που είχαμε λάβει σχετικές ε, διαβεβαιώσεις το 2005 δεν προέκυψε όμως τίποτα έκτοτε. Έχω την εντύπωση ότι σε ό,τι αφορά την πορεία των απαραίτητων αλλαγών δεν υπάρχει και μεγάλος ενθουσιασμός μεταξύ των κρατικών αρχών. Και αυτό το δημοψήφισμα που ανακοινώθηκε Ε, αν δεν πάει καλά, θα απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο το Κυρκυζιστάν από το δρόμο της δημοκρατίας. Ε, εμένα με απασχολεί σε ποιους μπορούμε να βασιζόμαστε εκεί. Θεωρώ ότι προ πενταετίας είχαμε υποτιμήσει την κατάσταση που διαμορφώθηκε στο Κυρκυζιστάν. Περιμέναμε περισσότερα Τώρα αντιμετωπίζουμε πάλι μια δοκιμασία. Είναι απαραίτητο να γίνουν προσπάθειες και είναι απαραίτητο η διεθνή κοινότητα να βοηθήσει το Ορκιγιστάν να σταθεί στα πόδια του και σε ό,τι αφορά τη χρηστή διοίκηση και τη σωστή λειτουργία της κυβέρνησης. Είναι μικρή μεν η χώρα αυτή, αλλά βλέπουμε ότι μπορεί να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει οι δράσεις μας να είναι καλά μελετημένες. Καλή επιτυχία λοιπόν στην προσπάθειά σας. Κύριε. Σας, σας ευχαριστούμε κύριε Πέτερ, λέει ο κύριος Βίγκινη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μορέλ για την παρουσίαση σας των εργασιών μέχρι τώρα των διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονται και πολλοί συνάδελφοι δυστυχώς ενώ είναι από τα κυριότερα θέματα που θα χρειαστεί να χειριστούμε στο άμεσο μέλλον. Έχω ορισμένε ερωτήσεις, διότι η αποτίμηση της κατάστασης στο Κυρζιστάν και το Ουσμπεκιστάν είναι καθαρή και σαφής, δεν έχουμε διαφορές εδώ. Θέλουμε να δούμε απλώς πώς θα στηρίξουμε καλύτερα το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ερωτώ, πώς εκτιμάτε την κατάσταση ως προς το εξής. Υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθούν όλα αυτά, να εξαχθούν και στις γειτονικές χώρες τα προβλήματα. Και δεύτερον, θεωρείτε ότι η τωρινή κυβέρνηση του Κυργιστάν είναι σε θέση να επαναφέρει τον έλεγχο και πώς βλέπετε την ιδέα της αποστολής μιας διεθνούς δύναμης επιβολής της τάξης εκεί. Μπορεί έτσι να δημιουργούνταν οι συνθήκες για την απαραίτητη σταθερότητα με επόμενη φάση τη συμφιλίωση, την τιμωρία των υπευθύνων, Και τέλος, το κυριότερο θέμα στο Ουσμπεκιστάν είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε το ανθρωπιστικό πρόβλημα. Πώς το βλέπετε λοιπόν μπορούν να το αντιμετωπίσουν το μεθοριακό τους πρόβλημα με το Κρυγκριστάν Λένε ότι υπάρχουν 100.000 πρόσφυγες ήδη. Πώς, τι πληροφορίες έχετε. Ξέρω ότι η Ένωση προσπαθεί κάτι να κάνει και όσο πιο γρήγορα μπορεί. Αλλά τι ακριβώς συμβαίνει επί τόπου. Γιατί μπορεί να έχετε καλύτερες πληροφορίες από μας. Στο... Ευχαριστούμε κύριε Βίγγενινγκ και κυρία Χάουταλα για τρία ολόκληρα λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ υπάρχουν μαθήματα που μπορεί να πάρει η Ένωση από αυτή την τραγωδία. Πρώτον, Χρειάζεται περιφερειακή προσέγγιση. Πρέπει να ζητήσουμε από το Ουσμπεκιστάν, το Καζαχστάν να κάνουν μία προσπάθεια για να λύσουν τα σοβαρά ανθρωπιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και βέβαια η περιφερειακή προσέγγιση χρειάζεται και παντού αλλού. Ντου. Δεύτερον, νομίζω ότι δεύτερο μάθημα είναι ότι επειδή υπήρχαν προειδοποιητικά σημεία για το τι θα συνέβαινε έχουμε εκεί αυτιά και μάτια αυτό ερωτώ πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί γιατί εκείνες είναι οι καταλληλότερες για να οικοδομήσουν γέφυρες και να καταλήξουν στη συμφιλίωση πάβοντας την κατάχρηση εξουσίας. Σήμερα διάβασα ότι η Διεθνής Αμνηστία ζητάει άμεση, άμεσο άνοιγμα των συνόρων με το Κυργιστάν. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάτι τέτοιο, για να ζητήσει να επιμείνει από τις αρχές του Ουσμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Κυργιστάν να ανοίξουν τα σύνορά τους σε όλους όσους πρέπει θέλουν να φύγουν και να του ζητήσει συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ για την προστασία των προσφύγων. Τρίτον, η Διεθνής Αμνηστία ζητάει από τις τρεις κυβερνήσεις επίσης συνεργασία με όλα τα διεθνή σώματα και υπηρεσίες του ΟΗΕ για τη χορήγηση της απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας και για να μπορέσει η πάτη αρμοστία του ΟΗΕ να αναλάβει την περίθαλψη των προσφύγων. Λοιπόν, πώς μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις, ε, λογικές, τα λογικά αυτά αιτήματα. Μπορεί η Ένωση με οποιονδήποτε τρόπο να αναβιώσει την ε, συνεργασία που είχε κάποτε στην περιοχή αυτή για την ε, διασφάλιση της συλλογική ασφαλείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Χάουταλα. Ο κύριος Αγκουράκης για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχήν να εκφράσω και εγώ την ε, λύπη μου για το ότι τόσοι λίγοι συνάδελφοι παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό και τραγικό γεγονός. Ε, πριν θέσω τρία ερωτήματα στον ε, ε δόκτρα, ε, τον κύριο Μορέλ, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να κάνω την εξή επισήμανση. Νομίζω ότι το πρόβλημα στο Κυργιστάν αναδεικνύει ε, πάρα πολύ καθαρά αυτό που αρκετό καιρό υποστηρίζω στην Επιτροπή σας, ότι δηλαδή βρισκόμαστε σε μια καινούρια κατάσταση όπου υπάρχει ένας μεγάλος ανοιχτός ανταγωνισμός μεγάλων υπεραλιστικών δυνάμεων για το θέμα της ενέργειας. Ε, στο Κυργιστάν δεν είναι, δεν είναι πια κανένα μυστικό, γνωρίζουμε, υπάρχουν Ηνωμένε Πολιτείε, υπάρχει Αμερικάνικη βάση στη χώρα αυτή, υπάρχει η προσπάθεια της Ρωσίας να ελέγξει μια κατάσταση, υπάρχει το κοντινό Αφγανιστάν, υπάρχει γενικά μια αστάθεια. Και με αυτή την έννοια θα συμφωνήσω απόλυτα και με σας κύριε Πρόεδρε και με τον ε, Δόκτωρ Μορέλ ότι η κατάσταση στη χώρα αυτή ε, απειλεί να οξύνει την αστάθεια που ούτως ή άλλως υπάρχει από εδώ απορρέει το πρώτο ερώτημά μου ε, στον ε, δόκτωρ Μορέλ. Ε, ποια είναι κατά τη γνώμη του η, αιτία της διένεξης της εθνοτικής στο Κυργιστάν. ποιος είναι ο λόγος. γιατί έγινε η διένεξη. Μας είπε ότι υπήρχε ένα προηγούμενο ή περισσότερα. Ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς, αν μπορεί να μας φωτίσει. Δεύτερο ζήτημα, πόσο η κατάσταση στο Κυργιστάν, κατά τη γνώμη του, συνδέεται με την αστάθεια στο Αφγανιστάν, η οποία σήμερα, από ό,τι όλοι διαβάσαμε και μάθαμε, οξύνεται ακόμα περισσότερο λόγω της διένεξης του Προέδρου Ομπάμα με τον διοικητή των ατοικών δυνάμεων στη χώρα αυτή. Τρίτη ερώτηση, και τελειώνω με αυτό, αναρωτιέμαι, ε, μάλλον ε, ε, πρώτη αναρωτιέμαι, κύριε Πρόεδρε, πόσο σωστό είναι να γίνουν οι εκλογές το άμεσο χρονικό διάστημα και πώς αυτές οι εκλογές θα νομοποιηθούν τη στιγμή που ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας απουσιάζει, δεν θα μπορεί καν να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Και τελειώνω με το εξής ερώτημα. Ε, αν υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί για τον αριθμό των ε, προσφύγων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, πώς είναι αυτή η περιπτώσει γενικά, ε, και εάν εκτιμούμε ότι θα επιστρέψουν όλοι. Γιατί διάβασα σε κάποιο, στο διεθνή τύπο, ότι πολλοί από αυτούς αρνούνται να επιστρέψουν γιατί φοβούνται ε, τις συνέπειες ε, για τη ζωή τους. Πολλοί από αυτούς σκέφτονται να μείνουν στο Ουσμπεκιστάν και αρκετοί μάλιστα γίνεται λόγος να, να πάνε στη Ρωσία. Πώς έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. για τρία λεπτά. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η κατάσταση στο Κυργιστάν ήταν προβλέψιμη διότι υπήρχαν ήδη, είχαν σημειωθεί ήδη πολλές διαμάχες εθνοτικές και δυστυχώς αυτό το αγνοήσαμε στην Ευρώπη. Θα ήθελα να μου πείτε αν η κατάσταση αυτή μπορεί μεσοπρόθεσμα να διορθωθεί δεδομένου του ότι διστάζει να παρέμβει η Ρωσία όπως το συνηθίζει όταν πρόκειται για σταθεροποίηση της περιοχής. Θεωρείται ότι μπορεί να υπάρξει πολιτική συνένεση για να ληφθεί κάποια απόφαση αποστολής ειρηνευτικής ή σταθεροποιητικής δύναμης εκεί και θεωρείται σωστό ή πρέπει η Ένωση να ζητήσει τη χρήση battle groups. Πώς βλέπετε την κατάσταση στο νότο της χώρας γύρω στην πόλη ως, διότι μερικοί μιλάνε για 800.000 πρόσφυγες, άλλοι για 100.000 αλλά φαίνεται ότι η ανθρωπιστική κατάσταση είναι πάντως σοβαρή και απαιτεί μια άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι η Πάτη εκπρόσωπος θα μπορούσε να, με αυτή την ευκαιρία να κάνει πιο ορατή την παρουσία της Ένωσης χορηγώντας μεταξύ άλλων και χρηματική βοήθεια. Τελευταίο ερώτημα Υπάρχει καμία πληροφορία για τον αριθμό των θυμάτων που προξένησε ο Κυργιζικός στρατός. Γιατί σύμφωνα με τις επίσημες εκθέσεις ο αριθμός τους είναι μικρός, αλλά υπάρχουν πηγές που μιλούν για 2.000 φωνευθέντες. Σας ευχαριστώ κύριε Νικολάη. Θα παρακαλέσουμε τον ε, δόκτωρα Μορέλ να λάβει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι για τις ερωτήσεις που θα μου επιτρέψουν να μπω σε κάπως περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέταση μιας καταστάσεως που θα μας απασχολήσει ακόμα για μέγα διάστημα. έχει περάσει τώρα και στην κοιλάδα Φεργάνα πέρα από την Μεθόριο και η κοιλάδα αυτή ήταν πάντοτε σημαντική, σημαντικό πέρασμα και με, ε, και με είχε σε ανάμειξη πληθυσμών αλλά επίσης είναι και το θέμα της ε, ε διανομής του νερού με κατασκευή ε, έργων, φραγμάτων Γενικά υπάρχουν λοιπόν πολλοί παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν κρίση και μιλισμονούμε και την γετνίαση με το Αφγανιστάν. Για τον κύριο λέει πρώτα. Πώς η χώρα αυτή δεν έχει ένα ενιαίο όραμα, ποιοι είναι οι σύμμαχοι, ποιοι είναι αυτοί που ε, συμμερίζονται το δικό μας πολιτικό όραμα. Ας είμαστε σαφείς. Υπάρχει πρώτα εγώ ήμουν ε, ήδη από το 1992 πρέσβης της Γαλλίας στο Κυρκιστάν ειδικά σε αυτή την μικρή χώρα η οποία ήθελε κατά κάποιο τρόπο να βλέπει τον εαυτό της ως Ελβετία της ε, Κεντρικής, ε, της Κεντρικής Ασίας. Υπήρχαν οι προσδοκίες ενός μικρού λαού ε, που περικλείεται από μεγάλες χώρες, μια προσπάθεια δηλαδή να βρει μια ταυτότητα. Έγινε μια έκκληση στην Ευρώπη που θυμούμε συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος τάσης. Ήταν μια προσπάθεια να βρεθούν κάποιες λύσεις για χώρες που ήταν μακρινές για μας, αλλά ήταν όμως χώρα η οποία ήταν γειτονική με την Κίνα, την οποία τη γνωρίζαμε ελάχιστα. Ε, κάναμε τέτοιες ε, προσπάθειες πάντως, ε, δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τους. Μία χώρα άνοιξε πρεσβεία τότε, ενώ υπάρχουν στο διπλανό Καζακστάν 15 και μία μόνο πλήρης ε, πρεσβεία στο Κυργιστάν, η γερμανική, με έναν εντεταλμένο Γάλλο. Και αυτό είναι όλο. Δύο. Συν τώρα μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πλήρους λειτουργίας, αλλά ακόμα βρίσκεται σε επίπεδο διαχειριστών προγραμμάτων, δεν είναι ακόμα πλήρως ε, λειτουργική. Δεν δέχθηκε λοιπόν η χώρα αυτή πλήρη ευρωπαϊκή παρουσία και αυτό έχει συνέπειες σε ό,τι αφορά την ανάληψη δράσεως επιτόπου. Βέβαια, του τουλεχθέντος σιγά σιγά τα προγράμματα αυτά αρχίζουν και ε, έχουν μια ευρύτερη βάση. Λειτουργεί η ε, Ευρώπη εκεί. Υπάρχουν περίπου 300.000 ε, άνθρωποι στο όριο της φτώχειας αλλά έχουν ένα εισόδημα μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και μια δεκαετία. Έχουμε λοιπόν καταφέρει αρκετά πράγματα για να συμβάλλουμε στη σταθεροποίηση της χώρας αυτής. Δεν είναι επαρκή, αλλά ποιος άλλος έχει τέτοια προγράμματα για το Κυρκιστάν. Τα λέω αυτά για να δείξω ότι υπήρξε μια σταδιακή αύξηση της ε, ευρωπαϊκής εμπλοκής, που είναι και πιο μεθοδική εδώ και 3,5 χρόνια. Δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες, θα λέω αυτά μόνο για να δείξω ότι κάνουμε προσπάθεια και σε ό,τι αφορά τις πολιτικές επιλογές, που είναι και ο πυρήνας των ερωτήσεων του κ. Πέτρελε, μετά από τις εμπειρίες της προεδρευόμενης, της προεδρικής μάλλον δημοκρατίας, η επιλογή των ε, κυργησίων δεν είναι υπέρ ενός κοινοβουλευτικού καθεστώτος. Το χρησιμοποιούν τον όρο αυτό για να διακριθούν, να δείξουν ότι θέλουν να λάβουν μια διαφορετική προσέγγιση μετά από δύο αποτυχίες του προεδρικού συστήματος θέλουν ένα είδος μεικτού καθεστώτος. Εννοώ δηλαδή ότι τονίζουν τον κοινοβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά μέσα στα πλαίσια του ε, παρόντος συντάγματος έχουν ε, εκλογεί το Πρόεδρο με καθολική ψηφοφορία. Αυτό που είναι σημαντικό για το σχέδιο αυτού συντάγματος είναι η αναζήτηση ενός συστήματος ισορροπιών και ελέγχων που να λειτουργεί. έχει την εξή αξία η επιλογή του κοινοβουλευτικού συστήματος. Έχουν δει κατ' επανάληψη κινήματα στους, στους δρόμους, τη δημιουργία μικρότερων κινημάτων περιφερειακού, ακόμα και οικογενειακού χαρακτήρα που δεν έχουν επιτρέψει να σταθεροποιηθεί ο πολιτικός διάλογος. Για να σταθεροποιηθεί ο διάλογος αυτό πρέπει να γίνει μέσα στα πλαίσια ενός κοινοβουλίου αυτός είναι ο λόγος της επιλογής αυτής και σε, στη βάση ενός αναλογικού συστήματος εκλογών με ένα κατόφλι και με εθνικά ψηφοδέλτια να περάσουν από τα 100 κόμματα σε 6-7 ώστε να επικεντρωθεί και περισσότερο ο πολιτικός διάλογος αυτή θεωρούμε ότι είναι και η επιλογή της προσωρινής κυβέρνησης και θα περάσει από ένα δημοψήφισμα. Η κυβέρνηση θέλει να διασφαλίσει τη δυνατότητα να διεξάγονται εκλογές σε ολόκληρη τη χώρα. Αβέβαια η εξέλιξη αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει προς τα εκεί κινείται η ε, κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Για τον κύριο Βιγγένιν, για το ρόλο του Ουσμπεκιστάν στην υποδοχή των προσφύγων. υπολογίζουμε σε τουλάχιστον 400.000 τους πρόσφυγες ή εκτοπισμένους που έχουν δηλαδή διέλθει τα σύνορα που είναι πιο κοντά γιατί Τζαλαλαμπάντ και Ως απέχουν λίγα χιλιόμετρα μόνο από τα σύνορα αφού είναι μία μία και μόνη κοιλάδα η οποία διακόπτεται από αυτό το παράξενο κάπως σύνορο. επομένως η κοιλάδα χωρίζεται ανάμεσα σε Ουσβεκιστάν, Κυρκιστάν και Τατζικιστάν. Υπάρχουν περίπου 10.000 110.000 ε, περίπου οι οποίοι δήλθαν τα σύνορα ορισμένοι έμειναν πίσω για να ε, προστατεύσουν ε, τις περιοχές τους και υπάρχουν περίπου 100.000 οι οποίοι έχουν παραμείνει λοιπόν ε, στο Ουσμπεκιστάν και περίπου 35.000 από το σύνολο των 400.000 δεν θα ε, κάνω πια διάκριση μεταξύ προσφύγων και εκτοπισμένων αλλά ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνηση ας πούμε και φαίνεται πως έχουν επιστρέψει. Μένουν περίπου 100.000 λοιπόν στο Ουσμπεκιστάν και 300.000 ακόμα που είναι μέσα στο Κυρκιστάν, αλλά όπως είπα εκτοπισμένοι από τις εστίες τους. Αυτό που ενδιαφέρει να επιστρέψουν το δυνατόν συντομότερο. Σε ό,τι αφορά την άμεση επίγουσα βοήθεια ε, διατροφής, ε, ύδατος κλπ. Αυτή έχει ασφαλιστεί λίγο πολύ. Έρχονται τα εφόδια δηλαδή οι προσπάθειες και των μη κρατικών οργανώσεων και της διεθνούς κοινότητας φαίνεται πως λειτουργούν ικανοποιητικά. Με καλή υποδοχή από πλευρά των ουσμπεκικών αρχών και με προσπάθεια να διατεθούν ε, στους απολύτες ε, τα ε, εφόδια. Ο ύπατος εκπρόσωπος ήταν παρόν στο Ουσμπεκιστάν και λειτουργεί μέσω UNICEF ή PNUD ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες επιτόπου. Πραγματικά πλήρως λειτουργική η κατάσταση αυτή. Επίσης ο Ερθρός Σταυρός μπορεί και λειτουργεί, οι ιατροί χωρίς σύνορα, άλλες οργανώσεις είναι όλοι παρόντες εκεί. Οι ανάγκες λοιπόν έχουν καθοριστεί καλά, οι δομές από πλευρά του Ουσμπεκιστάν, όπω είπα, είναι πλήρω λειτουργικέ και δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπήρξε κάποια στιγμή προσωρινό κλείσιμο των συνόρων γιατί είχαν ε, ξεπεράσει τι ε, δυνατότητες υποδοχής από πλευρά του Ουσμπεκιστάν. Αλλά άνοιξαν ξανά. Αυτά μπορώ να πω τώρα από πλευρά του Ουσμπεκιστάν. Τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα διότι έχει χάσει τον έλεγχο η δημόσια αρχή από πλευράς Κυργιστάν ως και Τζαλαλαμπάντ. Τα πράγματα επανέρχονται σιγά σιγά. Η κυβέρνηση ε, αναλαμβάνει πλέον ξανά ε, τη δυνατότητα η προσωρινή πρόεδρος ιδιαίτερα θαραλέα διεξάγει επισκέψεις στα νοσοκομεία, ε, στις γειτονιές με τα οδοφράγματα αυτά τα οποία έγιναν για λόγους αυτοάμυνας έχουν σχεδόν αποσυρθεί τουλάχιστον έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία άκουσα τα νέα σήμερα ότι στο Ως η κυκλοφορία είναι λίγο πολύ ομαλή τα λεωφορεία κυκλοφορούν δεν λέω ότι όλα είναι απολύτως ομαλά αλλά η ιδέα της επιστροφής στις αιστείες είναι πλέον μια ε, πραγματικότητα ορατή. Υπήρχε μια ερώτηση ακόμα, κύριε Πρόεδρε, σχετικά με την παρουσία μιας δύναμης σταθεροποίησης. Δεν βρισκόμαστε ακόμα εκεί, γιατί κάτι τέτοιο χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βλέπουμε πόσο προσεκτική είναι προκειμένου η Ρωσία. Εκεί που μπορούμε να δράσουμε εμεί αμέσω, δηλαδή πολιτική υποστήριξη, ανθρωπιστική ε, βοήθεια από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά μπορούμε να τα προσφέρουμε ευθύ αμέσω. στα πλαίσια του ΟΑΣΕ στην Βιέννη. Αυτά είναι τα στοιχεία που μπορώ να σας ε, προσφέρω ως απάντηση. Ευχαριστούμε, δόκτωρα Μορέλ. Οι Γκόμες και Παλέτσκιτς έχουν δύο λεπτά ο καθένας για μία τελευταία ερώτηση, αν μπορείτε να παραμείνετε μέχρι τις 12. Κύριε Πρέσβη, κατανοώ ότι είπατε ότι αυτή τη στιγμή ο ΑΣΕ θα πρέπει να παρέμβει μέσα στα πλαίσια μιας αποστολής. Σε αυτά τα πλαίσια τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έπρεπε να πιέσουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει μία αποστολή ασφαλείας όπου να δεσμευτεί και ο ΑΣΕ. Μαζί με τις γείτονες χώρες όπως ε, η Ρωσία. Γιατί θεωρείτε ότι η Ρωσία ήταν επιφυλακτική ή ανταποκρίθηκε εν μέρη στο αίτημα της προσωρινής Προέδρου του Κυργιστάν. Ως προς την Κίνα, ξέρω ότι η Κίνα ε, έκλεισε τα σύνορά της, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα ακόμα και ως προς τις οικονομικές συναλλαγές με το Κυργιστάν. Ποιος είναι ο ρόλος της ε, Κίνας και μακροχρόνια Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να βρούμε μία λύση μέσα στα πλαίσια των συνόρων του ε, συνοριακού καθεστώτος, γιατί τα σύνορα άλλαξαν υπέρ της Κίνας τα τελευταία χρόνια. Παλέτσκης, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας για τα τραγικά γεγονότα στο Κυρβιστάν. Πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν την σταθερότητα στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας, ιδιαίτερα στις γειτονικές χώρες Ουσμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Καζαχστάν και ποιος είναι ο ρόλος του ριζοσπαστικού Ισλάμ στα γεγονότα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Παλέτσκης οι απαντήσεις τώρα. Θα απαντήσω σύντομα στα δύο αυτά ερωτήματα. Για τον ΟΑΣΕ. Νομίζω ότι είπα ότι συνεργαζόμαστε με τον ειδικό, τους, με τον ειδικό εκπρόσωπο του ΟΗΕ ήταν ο Γιάνν Κούπης και τώρα είναι ο Γιάνν Τσακ με τον πρέσβη Καρατζάνοφ του ΟΑΣΕ και ο ίδιος με εντολή από τη Λέβη Άστον κατευθείαν. Υπάρχει λοιπόν συντονισμός από την αρχή. Πρώτη φορά συναντηθήκαμε τρεις μέρες μετά το δράμα στον Μπισκέκ και από τότε βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή. Δεν πρωταγωνιστεί ο μεν ή ο δε και οι τρεις μαζί προσπαθούμε να συντονιστούμε για να μην υπάρξουν επικαλύψεις που θα ήταν τραγικό και να μην λέει ο ένας το ένα και ο άλλος το άλλο. Ενώ έχουμε μπροστά μας μία τραγική κατάσταση πρέπει αφού συμμεριζόμαστε τις αναλύσεις να μιλάμε και με την ίδια φωνή. Ο καθένας βέβαια χρησιμοποιεί τα μέσα που διαθέτει στη διάθεσή του για να υπάρχει καλύτερη κατανομή των εργασιών. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή για την αστυνομία, για την ασφάλεια, για την ανάκτηση από την κυβέρνηση του ελέγχου των δυνάμεων ασφαλείας, ο συντομότερος δρόμος είναι ο ΑΣΕ, η ΟΑΣΕ. Ακόμα το μελετάμε βέβαια, αλλά αυτές τις μέρες θα αποφασιστεί ποιο, ποια ακριβώς θα είναι η στήριξη έχουμε 50 εμπειρογνώμονες περίπου και καμιά εκατοστή άλλους που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για, όχι για να δράσουν επιτόπου αλλά για να βοηθήσουν να συνοδεύσουν τον έλεγχο από την αστυνομία που είναι και χωροφυλακή εκεί. Γιατί όλες αυτές οι δυνάμεις ασφαλείας ε, τάχασαν από το δράμα. Υπήρξε μια απώλεια λοιπόν εξουσίας εκεί, ένα κενό, σχετικό κενό εξουσίας. Πολλοί αστυνομικοί σκοτώθηκαν βέβαια και από τα γεγονότα. Και όλα αυτά δημιούργησαν κάποια βεβαιότητα. Η επιστροφή αυτή λοιπόν στον πολιτικό έλεγχο ή του πολιτικού ελέγχου στηρίζεται από τον ΟΑΣΕ που φαίνεται το καταλληλότερο όργανο, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει και εκείνη στη συζητήση του ΑΣΕ για το τι πρέπει να γίνει. Η Ρωσία. Η κυρία Γκόμες ρώτησε γιατί η Ρωσία διστάζει. Καταρχήν Στη Ρωσική Ομοσπονδία, στην Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων Κρατών συζητήθηκε το θέμα και για να μην υπάρξει κάποια βία αντίδραση λαϊκής εκδίκησης που θα χειροτέρευε ακόμη περισσότερο τα πράγματα και θα αύξανε τον κίνδυνο εμφυλίου πολέμου. Ο πρόεδρος και ο κύριος Λουκασένκο της Λευκορωσίας ο πρόεδρος που είχε καταφύγει στη Λευκορωσία έκαναν βέβαια πιο βιές δηλώσεις αλλά τελικά η κυρία Ταμπάγεβα μετά από τη δεύτερη φάση της κρίσης και τις εθνοτικές εκρήξεις στο Νότο ζήτησε εκ μέρους της Ρωσίας από τον CSTO να οργανώσει τα πράγματα για να αποφευχθούν οι εξωτερικές απειλές αλλά δεν προβλέφθηκε τίποτα για την εσωτερική κρίση. Παρά την ανταλλαγή απόψεων λοιπόν τελικά αποφάσισε η Ρωσία να απόσχει από οποιαδήποτε δράση. Η Κίνα και αυτή παρέμεινε αρκετά σιωπηλή. Ήδη από τις 7 Απριλίου στις κινήσεις μεταξύ των κινήσεων του Όχλου έγιναν επιθέσεις κατά της περιουσίας του Μπακίεφ Ε, λόγω βέβαια της, των αισθημάτων εκδίκησης που κυριαρχούσαν η εκδικητικότητα. Και στο Νότο και εκεί ήταν παρόσα η Κίνα, έκανε προσπάθειες να προστατεύσει τους πολίτες της. 1300 Κινέζοι μεταφέρθηκαν από την ΟΣ, πράγμα που δείχνει πόσο πολλοί ήταν παρόντες. Δεν έκλεισαν τα σύνορα με την Κίνα, απλώς πάγωσαν οι εμπορικές συναλλαγές που συνεισέφεραν κατά πολύ στην ευημερία της περιοχής και της κοιλάδας της Φεργάνα. Αυτά μπορούσα να σας πω. Τώρα για το ερώτημα του κυρίου Παλέτσκι για τους γείτονε. Το Καζαχστάν προσπάθησε να παίξει κάποιο ρόλο ως γείτονας αλλά και ως προεδρεύων σαν χώρα στον ΟΑΣΕ και υπήρξε επομένως ενεργό. Ήταν ένας από τους τρεις απεσταλμένους επιτόπου αλλά ταυτόχρονα φοβούμενο τη γενίκευση της Σύραξης έκλεισε τα σύνορά του. Τα καζαχοκυριχιζικά σύνορα είναι κλειστά και μερικώς άνοιξαν τουλάχιστον για τις τρέχουσες εμπορικές συναλλαγές. Δεν λύθηκε ακόμη αυτό και παραμένει δύσκολο. Για το Σμπεκιστάν τα σύνορα ελέγχονται, επιτρέπεται η διέλευση προσφύγων και η επιστροφή τους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι Ουσμπέκοι εμπόδισαν συμπατριώτες τους να περάσουν τα σύνορα για να πάνε να συμβάλλουν στην, να βοηθήσουν τους μειονοτικούς Ουσμπέκους που ζούσαν εκεί. Όσο για το Τατζικιστάν, εκεί δεν σημειώθηκε καμία ιδιαίτερη ένταση, αλλά ξέρουμε ότι από το Τατζικιστάν έρχονται αποσταθεροποιητικά και ακραία στοιχεία στο Κυργίσταν που έχουν τη λογική του ανταρτοπολέμου ή του Ισλαμισμού. Στο Βαζιριστάν ιδίω έχουν καταφύγει τέτοια στοιχεία σε συνεργασία με τους Ταλιμπάν χρησιμοποιώντας τους διαδρόμους του λαθρεμπορίου ναρκωτικών με τη γνωστή μέθοδο ναρκωτικά έναντι Και είναι και αυτό αποσταθεροποιητικός παράγοντας και για τις δύο γειτονικέ χώρες, Τατζικιστάν και Κυργιστάν. Δηλαδή, για να συνοψίσω, θα έλεγα ότι η δύσκολη κοινωνική κατάσταση του Κυρκυστάν. Η αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης και οι επιπτώσεις της αφγανικής διαμάχης είτε από κρέα στοιχεία, εξτρεμιστικά στοιχεία είτε μέσω των ναρκωτικών είναι σοβαρά στοιχεία που συνδυάστηκαν όλα σε αυτή την περίπτωση στην, ως και στην Τζελαλαμπάντα και εκεί πρέπει να γίνει και η προσπάθεια. Η διεθνής βοήθεια υπάρχει όμως και μπορούμε να μιλήσουμε ήδη για αναδόμηση και συμφιλίωση γιατί μόνο έτσι μπορούν να αποφευχθούν και χειρότερα. Είναι δύσκολα τα πράγματα αλλά ακόμη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μόνιμη συνεργασία με άλλους εταίρους και τις οργανώσεις που ανέφερα παίζει το ρόλο της και νομίζουμε ότι ο ρόλος αυτός ε, λήφθη, πραγματοποιήθηκε, δηλαδή κάναμε αυτό ακριβώς που έπρεπε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εισήγηση αυτή, πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση. Είδαμε πώς έχουν οι δραματικές εξελίξεις στην περιοχή, αλλά υπάρχει και κάποιο φως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρέσβη Μπακτιάρ Κούλιαμόφ που είναι μαζί μας. Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να σας δώσω το λόγο, αλλά θα μας διαβιβάσετε ένα γραπτό κείμενο για να δούμε τις, ε, δύσκολες, ε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ως προς τις, ε, τους πρόσφυγες που ανέρχονται σε 400.000 και οι οποίοι έχουν προσφύγει στη γειτονική χώρα. Θα προσπαθήσουμε να καταπραίνουμε τουλάχιστον, να ελαφρύνουμε την κατάσταση ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια και μετά θα συνεδριάσει το Διευρυμένο Προεδρείο. Σε τρία-τέσσερα λεπτά συνεχίζουμε.